Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, να αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Προτείνω έχετε δει την ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε παρατηρήσει, θεωρείτε εγκεκριμένη. Ανακοινώσει του Προέδρου. Ω συνήθω, σα έχουν κοινοποιηθεί οι γλώσσε για τι οποίε υπάρχει διερμηνία είναι οι γλώσσες των μελών της Επιτροπής Τάξε 2 και των προσκεκλημένων που χαιρετίζω. Θα τους ε, υποδεχτώ ως λίγο. Στα πλαίσια του Paper Smart δεν έχετε έγγραφα. Ηλεκτρονικά σας έχουν διανεμηθεί όλα τα πετούμενα έγγραφα. Αλλά φυσικά μπορείτε να εκτυπώσετε αυτά τα έγγραφα. Είναι ανοιχτή η συνεδρίαση για τους δημοσιογράφους και όλους όσους ε, ενδιαφέρονται να την παρακολουθήσουν τη σημερινή μας συνεδρίαση και να μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Όπως σας είχα πει το, την περασμένη εβδομάδα, ε, τα έγγραφα της Επιτροπής Κώδικα Διοντολογίας του Συμβουλίου είναι στη διάθεση όλων των μελών της Επιτροπής τάξε 2 και του επιτελείου του προσωπικού τους. σε μία αίθουσα στο Square de 10 ε, μέτρα από τη γραμματεία της Επιτροπής μας. 9 με 12.30 και 1.30 με 5.30 Δευτέρα με 5.00 και μέχρι τις 12.30 την Παρασκευή. Ώρες γραφείου δηλαδή. Ε, να κλείστε ραντεβού. Θα σας έλεγα, το έχουν κάνει ήδη κάποιοι. Ε, επικοινωνήστε με την γραμματεία, ούτως ώστε να έχετε πρόσβαση στα έγγραφα όταν τα χρειάζεστε. Φτάνουμε τώρα στο τρίτο σημείο της διάταξη, το πιο σημαντικό, ανταλλαγή απόψε με διάφορες ευρωπαϊκές τράπεζες. Οι συντονιστέ της Επιτροπή. θέλησαν, επειδή είναι αυξημένο ο αριθμό των προσκεκλημένων, να κάνουμε δύο διαφορετικέ συνεδριάσει για τους εκπροσώπους των τραπεζών, για τις ακροάσει δηλαδή. Ε, και ε, ανάλογα με τα στοιχεία του ενεργητικού, ανάλογα με το μέγεθος των ε, τραπεζών αυτών, βάσει των στοιχείων της ΕΚΤ, ταξινομήθηκαν σε δύο κατηγορίες. Ο στόχος είναι να διαπιστώσουμε ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν στην, στην πολιτική φορολογικού σχεδιασμού των πελατών τους και κυρίως των πελατών που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς μας και ενδιαφερόντων μας, δηλαδή των πολυεθνικών διότι οι τράπεζες εξορισμού ε, συνοδεύουν όλες τις κινήσεις ε, των πελατών τους, είναι ούτως ή άλλως πολυεθνικές ε, οντότητες, διαθέτουν ένα ευρύτατο φάσμα χρηματοπιστωτικών προϊόντων που την χάνουν διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με το κράτο μέλο, τα υβριδικά επωνομαζόμενα προϊόντα και μπορούν να προσφέρουν στου πελάτε του υπηρεσίες φορολογικής διερεύνησης όπως το διαπιστώσαμε την περασμένη εβδομάδα στις ακροάσεις που κάναμε ε, για διάφορες πολυεθνικές. Φερμπίν, ε, για να υποφελθούν από το σύστημα της μετατόπισης της φορολόγησης, το περίφημο αμερικανικό deferral, το ε, κρατούσα στα ζεστά τα, τα χρήματα σε κάποια νησιά μη επαναπατρίζοντας ε, όλα τα κέρδη λοιπόν ε, στη ΣΥΠΑ ελπίζοντας ε, ότι για μεγάλη χρονική περίοδο οι ΕΣΑΗ θα διαφύγουν από την καταβολή των φόρων στη ΣΥΠΑ. Θα δούμε λοιπόν τις εμπειρίες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών σήμερα και καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε για την παρουσία τους στους εκπροσώπους Κρετή Αγκρικόλ και της e ΕΝΖ που θα είναι στο πρώτο πάνελ, Νόρτεα επίσης Σαντάντερ, δεύτερο πάνελ, UBS και Unicredit, τρίτο πάνελ. Έχουμε επίσης τη συμφωνία επί της αρχής ούτως ώστε στις 4 Απριλίου στην επόμενη συνεδρίασή μας να έρθει η Deutsche Bank και η Royal Bank of Scotland. Μέσα στο ίδιο πνεύμα, μέσα στο ίδιο πλαίσιο τους προσκαλούμε. Είναι οι σημαντικότερες τράπεζες που έχουν την έδρα τους σε διαφορετικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρόπο ώστε να σχηματίσουμε μια ε, όσο το δυνατόν πιο σφαιρική και ε, πλήρη εικόνα ε, μπορούμε. Όπως και την περασμένη εβδομάδα με τις πολυεθνικές. Μετά από μία αρχική γραμμική παρουσίαση που σας προτείνω να περιορίσουμε σε ένα πεντάλεπτο, θα ακούσουμε τους εκπροσώπους της Κρέδια Γκρικόλ και της e για πέντε λεπτά έκαστος και μετά κλασική σειρά ερωταπαντήσεων όπως και στα πάνελ της περασμένης εβδομάδας, είναι δυνατόν ε, οι ομιλητές να θέλουν να απευθύνουν το ερώτημά τους σε έναν από τους δύο προσκεκλημένους, σε έναν από τους προσκεκλημένους ή και στους δύο. Όπως λοιπόν και την περασμένη εβδομάδα, επειδή λειτουργήσε σύρως το σύστημα, εάν ε, απευθύνεται το ερώτημα σε ένα μόνο προσκεκλημένο, σε μία τράπεζα, τότε έχουμε τα σλότ πέντε λεπτά για την ερώτηση και την απάντηση, δύο για την ερώτηση και τρία για την απάντηση, χοντρικά. Εάν τώρα ο, ο θέλει να υποβάλει το ερώτημα και στους δύο προσκεκλημένους, είτε για να θέσει το ίδιο ερώτημα, είτε για διαφορετικά ερωτήματα, τότε έχουμε δύο χρονοθυρίδες τρίλεπτες. Μία, ένα λεπτό για την ερώτηση, ε, τρία για την απάντηση ε, για την ε, πρώτη και για τη δεύτερη μετά τράπεζα. Ο Jean-Claude Μπαλάτ, Διευθυντής Επιχειρήσεων της Κρετή θα πάρει το λόγο για πέντε λεπτά. Κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, με ο Ζωζάν Σαλ ε, Μπαρελά. Δεν είμαι διευθυντή των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, αλλά των φορολογικών υποθέσεων τη Credit Αγκρικόλ ε, SA, ανώνυμης εταιρεία, ε, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και είναι το βασικό όργανο τη Credit Αγκρικόλ. Τι σημαίνει αυτό. Βάση του νόμου και είναι ο νομισματικό και χρηματοπιστωτικό γαλλικό κώδικα, μεριμνούμε ώστε στο εσωτερικό του ομίλου και τηρώντα την νομοθεσία με όλες τις δομές του Κρεντή Αγκρικόλα που συνδέονται με την κεντρική δομή να παρακολουθούμε τις δραστηριότητες όλων των οντοτήτων. Είμαστε ο πρώτος χρηματοδότης της γαλλικής οικονομίας και της, ε, του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη. Έχουμε σχέσεις με το retail banking, τις ε, τράπεζες ε, των καταναλωτών δηλαδή. Εκπροσωπούμε τράπεζες με, με στοιχεία ενεργετικού για τις μεγάλες επιχειρήσεις όπως η Αναντή και είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων. Ε, λειτουργούμε σε συνεργατική βάση, βάση αμοιβιοποίηση, σε 9 εκατομμύρια μέτοχοι, 1 ε, εκατομμύριο για την εκρατεία Γκρικόλ ΕΣΑ, που είναι η εταιρεία που έχει τους περισσότερους μετόχους ε, στη Γαλλία, 52 εκατομμύρια πελάτες και 140.000 συνεργάτες. Το ε, είμαστε μια καθολική τράπεζα εγκύτητας, ε, δηλαδή υπάρχει, ε, έχουμε τα αποταμιευτήρια στη Γαλλία που είναι οι βασικές εταιρείε μας στην Γαλλία αλλά και στην Ιταλία έχουμε υποκαταστήματα, έχουμε διάφορα υποκαταστήματα που ασχολούνται με την τραπεζική, την καταναλωτική συγγνώμη πίστη, την τιμολόγηση, τη χρηματοδότηση, τις επενδύσεις, είναι ευρύ το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Σε 33 χώρες έχουμε παρουσία. Ως επιτοπλίστων όμως δραστηριοποιούμαστε στη Γαλλία ε, και το 75% του ισολογισμού μας ως εκ τούτου έρχεται από την Γαλλία και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, λειτουργούμε ως επιτοπλίστων για τα προϊόντα μας διότι πέρα από τη Γαλλία στην Ιταλία έχουμε χιλιά υποκαταστήματα αλλά και στην Πολωνία έχουμε πάνω από 400 υποκαταστήματα. Αυτή η δραστηριότητα ε, φαίνεται από τους φόρους που πληρώνει ο Όμιλος ε, στην Γαλλία, στο γαλλικό κράτος ε, πέρα από το 2,3 δισεκατομμύρια που πληρώνουμε σε εισφορές, 5 δις φόρους καταβάλουμε επίσης, εκ των οποίων 2,2 για εταιρικό φόρο στη Γαλλία το 2015, 600 εκατομμύρια φόρους για τους μισθούς και ε, έχουμε τον φόρο παραγωγής και δεν ε, μας επιστρέφεται ο ΦΠΑ. Επίσης ε, πληρώνουμε λίγο παραπάνω από ένα δις ε, ε, σε φόρους προς τις διάφορες διοικητικές αρχές των κρατών όπου έχουμε υποκαταστήματα. Για το 2015 σε επίπεδο ομίλου ο συνολικός ουσιαστικός φορολογικός συντελεστής είναι 33,3% είναι ιδιαίτερα υψηλός όμως υπενθυμίζω ότι και πάλι ως επιτοπλίστων δραστηριοποιούμαστε στη Γαλλία μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 ήταν στο 38%. Ε, τώρα, για το κρατή ακρικολ, κάνουμε στο φορολογικό τομέα. Σε ολόκληρο τον κόσμο ε, προσφέρουμε υπηρεσίες ε, και έχουμε 100 περίπου εργαζόμενους. Ε, κυρίως στη Γαλλία δουλεύουν, αλλά έχουμε και κάποιους στην Ιταλία, στο Λονδίνο και στην Νέα Υόρκη, αλλά και στην Ασία. Οι φοροτεχνικοί αυτοί λοιπόν ασχολούνται κυρίως με ε, τον, τον ίδιο το όμιλο, δηλαδή φορολογική δήλωση, παρακολούθηση, διαχείριση του φορολογικού βάρους. Ε, αντίθετα, ποτέ ε, δεν προσφέρουμε φορολογικές υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών προς τους πελάτες μας. Αυτό απαγορεύεται διότι στη Γαλλία όπως και σε πολλές άλλες χώρες, υπάρχει ένα μονοπόλιο για την άσκηση αυτού του δικαιώματος και το διαθέτουν μόνο οι φορολογικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι. ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα απαγορεύεται να παρέχουμε τέτοιες υπηρεσίες πέραν από αυτές που είναι συναφείς προς τα επενδυτικά μας ε, τραπεζικά προϊόντα. Παραδείγματος χάρη για απλά προϊόντα που οδηγούν σε φορολογικές εκπτώσεις και απευθυνόμαστε κυρίως σε ιδιώτες. Όταν ε, κάνει συναλλαγές ε, περίπλοκες ο ιδιώτης πρέπει να γίνουν αποδεκτές και να εγκριθούν από τις επιτροπές αρμόδιες για αυτά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που έχουμε στον όμιλό μας υπό την ευθύνη κυρίως της Γενικής Διεύθυνσης Συμβατότητας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικού Σχεδιασμού που έχουν δικαίωμα βέτο σε σχέση με τα προϊόντα. Νομίζω ότι εξέπνευσε ο χρόνος μου. Ε, πρόεδρε, ειδού εν ολίγης, ε, ποιο είναι το πλαίσιο δραστηριοτήτων της Κρεντή Αγκρικόλους προς τα φορολογικά ζητήματα. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Ζητώ συγγνώμη που έκανα λάθος και για το όνομά ε, σας και για την ιδιότητά σας. Θα δώσω τώρα το λόγο και πάλι για πέντε λεπτά στον κύριο Σκίπερ που είναι ο φορολογικός διευθυντής του ομίλου ING για πέντε λεπτά επίσης. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση στην ακρόαση αυτή της ειδική Υποεπιτροπής ε, για τις φορολογικές αποφάσεις. Ρόμ Χίπερ λέγομαι και είμαι αρμόδιος για θέματα φορολογικά σε παγκόσμιο επίπεδο στην ING από το 2014. Να σας κάνουμε εισαγωγή. Η ING είναι μια τράπεζα που λειτουργεί παγκοσμίω σε ελιανική τραπεζική, σε πάνω από 40 χώρες με έδρα στο Μπενελούξ. Γύρω στο 80% των 58.000 θέσεων εργασίας ε, που έχουμε, αλλά και των πελατών λιανικής, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να αφαιρθώ σε τρία θέματα. Την προσέγγισή μας στα φορολογικά, την προσέγγισή μας ε, στα φορολογικά των πελατών μας, τις συστάσεις μας ε, για ένα αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο. Πρώτο θέμα, η ING ακολουθεί μια συνετή προσέγγιση όσον αφορά τα φορολογικά. Όσον αφορά λοιπόν τους δικούς μας φόρους σημαίνει πως ο φόρος ακολουθεί την δουλειά μας και όχι το αντίστροφο. Ξεκινάμε λοιπόν από ένα οικονομικό σκεπτικό, οπότε δεν ακολουθούμε μόνο το γράμμα του νόμου αλλά και το πνεύμα του νόμου για τις φορολογικές αποφάσεις. Η προσέγγιση μας αυτή φαίνεται από το ότι πληρώνουμε παγκοσμίως ένα φορολογικό συντελεστή 26% πλην των άλλων ε, φορολογικών ε, τραπεζικών φόρων που πληρώνουμε σε πολλές χώρες, σε διάφορες ε, τράπεζες. Εάν λοιπόν αθροίσουμε τους τραπεζικούς και τους εταιρικούς φόρους, το συνολικό φορολογικό βάρος στα κέρδη μας είναι πάνω από 40%. Η προσέγγισή μας επίσης φαίνεται και από τις συστάσεις αναχώρα που συμπεριλαμβάνουμε στους ε, ετήσιους λογαριασμούς μας από το 2014 σύμφωνα με τις απαιτήσεις οδηγίας CRD4. Από εκεί πέρα συμπεραίνουμε πως τα οικονομικά μας αποτελέσματα αναφέρονται και φορολογούνται σε, με τοπικούς συντελεστές στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε. Για να καταλήξω λοιπόν. Και οι πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές ε, και οι ε, εκθέσεις αναχώρα δείχνουν πως οι φόροι πληρώνονται εκεί πέρα που δημιουργείται η αξία. Δεύτερον, όσον αφορά την σημερινή ακρόαση θα ήθελα να εξηγήσω τα εξή για την θέση μας για την φορολογία των πελατών μας. Πριν ε, το κάνω όμως θα ήθελα να σημειώσω το εξή. Όποιον ρόλο έχει μια τράπεζα στα φορολογικά των πελατών, οι, τράπεζα, οι πελάτες είναι πάντα υπεύθυνοι για τα δικά Για να επανέλθουμε λοιπόν στην θέση μας για τα φορολογικά των πελατών μας. Πρώτα απ' όλα, από σκοπιά πολιτικής, ε, εμείς ε, δεν δίνουμε φορολογικές σύμβουλες. Αυτό υπάρχει και στις φορολογικές αρχές μας που είναι δημόσιες και ο λόγος είναι πως ε, η βασική μας δραστηριότητα είναι τραπεζικές και όχι φορολογικές υπηρεσίες. Εμείς κάνουμε συναλλαγές με τους ε, πελάτες μας ή για λόγους επιχειρηματικούς όχι φορολογικούς. Δεύτερον, στηρίζουμε τις ε, φορολογικές αρχές τις προσπάθειές τους ε, να συλλάβουν την φοροδιαφυγή με το να συμμετέχουμε στις πρωτοβουλίες αυτόματος ανταλλαγής προφοριών όπως η ΦΑΤΚΑ και η ΣΥΑΡΕΣ. Με άλλα λόγια δίνουμε στις φορολογικές αρχές πληροφορίες για τους πελάτες μας για να μπορούν μετά οι αρχές να ελέγχουν αν συμμορφώνονται αυτοί ως φορολογούμενοι τρίτο και τελευταίο. Θέλαμε να σημειώσουμε πως ένα αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο για τη φορολογία, ιδεοδό σε παγκόσμιο πλαίσιο, είναι μια σωστή αφετηρία για να είμαστε αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της επιθετικής φοροαποφυγής. Γι' αυτό θεωρούμε πως το BEPS και η οδηγία κατά της φοροαποφυγής είναι σημαντικά βήματα σε σωστή κατεύθυνση. Όμως, θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ σημαντική να μην καταλήξουν αυτές τις προσπάθειες σε διπλή φορολογία και να διασφαλιστεί η ανταγωνιστική θέση της Ευρώπης. Καλωσορίζουμε λοιπόν το σημαντικό έργο της Επιτροπής αυτής και της ε, Κομισιόν. Ευχαρίστως να επεκταθώ στην ανταλλαγή απόψε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και τους δύο που παρουσιάσατε πολύ ωραία και συνοπτικά στον χρόνο που σας είχε οριστεί τις δραστηριότητες των ομίλων σας. Και τώρα έχουμε την κυρία Χούμπνερ, εξ ονόματος του ΕΛΚΑ. Αντανούτα, σε ποιον απευθύνεις τα ερωτήματα, τι θέλετε να πω. Τότε θα κάνω και τις δύο ερωτήσεις μαζί. Λοιπόν, για το θέμα που σχετίζεται με αυτό το νέο σύμπαν στο οποίο όλοι είμαστε αναμειγμένοι για αυτή τη βαθύτερη και ευρύτερη ανταλλαγή πληροφοριών που αποτελεί ένα νέο στάνταρ στην Ευρώπη και Θέλουμε να ξέρουμε, εσείς είστε υπεύθυνοι για αυτές τις ανταλλαγές πληροφοριών και πρέπει να ανακοινώνετε και τις αντίστοιχες, κοινοποιείτε μάλλον τις αντίστοιχες πληροφορίες σε αρμόδιες αρχές, καθώς και τα έσοδα που καλύπτονται από την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία και την νομοθεσία κατά του ξεπλήματος χρήματος. Εσείς ως τράπεζες λοιπόν είσαστε μέσα στην αλυσίδα πληροφόρησης που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε παράνομες συμπεριφορές αλλά και να εξασφαλίσουμε το συντονισμό ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Αρχές των διαφορών χωρών. Το ερώτημά μου αφορά την πείρα σας, αλλά και την αντίληψή σας για αυτή τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, μπορούν ε, κατά τη γνώμη σας οι τράπεζες και οι μεγάλες τράπεζες της, της Ευρώπης να συμβαδίσουν ε, με όλες αυτές τις εξελίξεις, μπορούν να σταθούν στο ύψος ε, των προκλήσεων της αναδιοργάνωσης που επιφέρει σημαντικό κόστος η προσαρμογή σε αυτές τις νέες προδιαγραφές. Υπάρχουν κάποιες καλύτερες πρακτικές σε σχέση με τα όσα κάνετε την τελευταία περίοδο. Και επίσης ποια είναι η γνώμη σας για τη συνεχιζόμενη τυποποίηση των δεδομένων, ας πούμε, για τον αριθμό ε, ταυτότητα, του ταυτότητα του Ευρωπαίου Φορολογούμενου που πιέζουμε εδώ και αρκετό καιρό εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ποια είναι λοιπόν η ε, αντίληψή σας για αυτή τη νέα περίοδο ανταλλαγή ανταλλαγής πληροφοριών μέσα σε αυτό το πλαίσιο προκλήσεων. Και να θέσω και τη δεύτερη μου ερώτηση. Όχι, εντάξει. Εσείς αποφασίζετε, εσείς σας το είπα από την αρχή. Είναι η ίδια ερώτηση και για τους δυο ομιλητές. Ναι. Παρακαλώ, δύο λεπτά και δύο λεπτά έκαστος. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Καταρχάς, όπως είπα και στην αρχική μου δήλωση, Υποστηρίζουμε πλήρως την, ε, τις ε, πρωτοβουλίες ε, ανταλλαγής πληροφοριών όπως το CRS και το, και το Και θεωρούμε πως οι, μέθοδες, οι μέθοδοι αυτές βοηθούν. Το CRS είναι καλό παράδειγμα γιατί πήρε την πρωτοβουλία της ΒΑΤΚΑ και έφτιαξε μια τελείως νέα προσέγγιση, οπότε για τις τράπεζες, αν και η ΦΑΤΚΑ και οι CRS Ε, απαιτούν αρκετή δουλειά για να εφαρμοστούν από πλευρά των τραπεζών γιατί έχουμε να κάνουμε με αλλαγές στα συστήματα στις επιχειρήσεις, στις επιχειρήσεις μας, στις διαδικασίες μας αλλά όσο περισσότερο το διατηρούμε τυποποιημένο είναι προς όφελος όλων μας. Ελπίζω ότι απάντησα στην ερώτησή σας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαλά. από την Κρεντή Αγκρικόλ. απόλυτα τα όσα είπε ο συνάδελφος. Να προσθέσω ότι δεν είναι νέο οι τράπεζες να χρησιμοποιούνται ώστε να δίνουν πληροφορίες. Εδώ και χρόνια, ξέρετε, για παράδειγμα στην Γαλλία, δίνουμε τις πληροφορίες στην φορολογική μας αρχή για να τον υπολογισμό των ε, ε, εισοδημάτων. Η ΦΑΤΚΑ και οι CRS ε, έχουν ξεκινήσει την, ανταλλαγή, την αυτόματη ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών. Είναι βέβαια ένα τυποποιημένο και ρυθμισμένο πλαίσιο και φυσικά και το εφαρμόζουμε και βεβαίως ήταν σημαντικό το κόστος εφαρμογής, αλλά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι όντως μπαίνουμε σε νέα εποχή. Και απόδειξη είναι ότι στον προγραμματισμό των μεσοπρόθεσμων του ομίλου μου ανακοίνωσε ο όμιλος ότι ένα δις ευρώ θα αφιερωθεί στις λειτουργίες συμμόρφωση και κίνδυνος. Ναι, ακριβώς ε, ε, είμαστε σε θέση και ετοιμαζόμαστε για να δίνουμε τις πληροφορίες που μας ζητώνται. Μα δεν είναι όμως κάτι νέο, επαναλαμβάνω. Επεταχύνεται το, η διαδικασία, αλλά δεν είναι κάτι νέο. Μάλιστα. Από πλευρά των σοσιαλιστών δίνω το λόγο στον Γιέπε Κόφουτ που είναι και εισηγητής. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τις τράπεζες που ήρθαν εδώ. Πρώτα απ' όλα κάνω μία ερώτηση στην Credit ε, Εγκρικόλ. Πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα να ακούσω από σας. Έχετε υπογράψει κάποιες ε, φορολογικές ρυθμίσεις με τις αρχές στο Λουξεμβούργο. Και αν μπορείτε επίσης να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες για την έκθεση της προηγούμενης εβδομάδας ε, της Oxfam που έδειξε πως ε, ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής σας στην Ιρλανδία ήταν μόλις 4% και λέτε πως ε, δεν έχετε λάβει δημοσία κονδύλια από την Ιρλανδία, αλλά τότε πώς βγαίνει τόσο χαμηλός πραγματικός φορολογικός και προς την Credit Agricole. Έχετε θηγατρικές ε, στα Virgin Islands ή έκλεισαν όπως είχατε πει. Μετά για την ING διάβασα μια έκθεση του Σεπτεμβρίου 2014 πως έχετε επενδυτικά ταμεία στα Cayman στις νήσους ε, Κέιμαν. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αν έχουν δοθεί δάνεια σε οχήματα ειδικής, ειδικού σκοπού όπως ανέφερε η έκθεση που προανέφερα και για τους δύο σας υπό το καθεστώς των εκθέσεων αναχώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω θεωρείτε πως είναι κάτι το χρήσιμο για την αύξηση της ε, διαφάνειας και θα έπρεπε να ισχύει σε όλες τις, για όλες τις πολυεθνικές εταιρείες και όχι μόνο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δύο λεπτά για την Credit Agricole και άλλα δύο για την ING. Κύριε, Κύριε Διευθυντά, όσον αφορά τις διάφορες χώρες που παραθέσατε, όντως εδώ και τρία χρόνια δημοσιεύουμε και αυτό συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια μας ε, έκθεση έκθεσης ανά χώρα. Και προφανώς είναι γνωστό αυτό για όλους. Μάλιστα, είμαστε και στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για μια σημαντική ε, χρηματοπιστωτική ε, κέντρο και ε, δύο θηγατρικές μας έχουν υπογράψει δύο ειδικέ ε, φορολογικές ρυθμίσεις με το Λουξεμβούργο. Όσον αφορά την Ιρλανδία, να θυμίσω ότι το ποσοστό φορολόγησης στις εταιρείες είναι 12,5% και αν ο φόρτος ο φορολογικός που φαίνεται στην ετήσια μας έκθεση είναι σχετικά μικρός, αυτό οφείλεται ε, στην ιδιαιτερότητα της Ιρλανδίας ότι δηλαδή φιλοξενεί διάφορα ασφαλιστικά ταμεία που είναι διαφανείς δομές. Το αποτέλεσμα αυτών ε, περιλαμβάνεται στις εκθέσεις αλλά η φορολόγησή τους γίνεται σε επίπεδο του ε, συνδεδεμένου μέλους, ο οποίος πληρώνει ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση το φόρο του στην Γαλλία. Πρόκειται για την ΑΣΕΚΑ. Ε, Τώρα, έχουμε 4 ή 5, αν θυμάμαι καλά, δομές ε, ε, ιδιωτικής, ε, ιδιωτικές τράπεζες στα Virgin Islands που έχουν κλείσει τώρα και νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τις, τα τρία αυτά καταστήματα και ολοκληρώνονται όπου να είναι και για τα υπόλοιπα δύο. Ευχαριστώ, κύριο Σίφερ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ για τις ε, εκθέσεις ε, αναχώρα. Στηρίζουμε πλήρως ε, το σύστημα αυτό. Θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να αυξηθεί η διαφάνεια για όλους τους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να δούμε τους φορολογικούς κινδύνους. Και τέλος θεωρούμε πως επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ διαφάνειας ε, και αποκάλυψης εταιρικών πληροφοριών. Και αυτό είναι σημαντικό. Και αν δείτε τις δηλώσεις αναχώρα της ε, ING αποδεικνύουν το ότι πληρώνουμε φόρους ε, στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε. Και εκεί όπου δημιουργείται η πραγματική εταιρική αξία δύο πολύ σημαντικές αρχές για εμάς. Για την δεύτερη ερώτησή σας, οι οντότητες ε, στις οποίες ε, αναφερθήκατε ε, υπάρχουν, αλλά για επιχειρηματικούς, όχι για φορολογικούς λόγους. Δεν κρύβουμε κέρδη εκεί και αυτό φαίνεται και στις εκθέσεις που προανέφερα. Ε, θα τα βρείτε αυτά στις ε, εκθέσεις και φαίνεται εκεί πέρα ποια είναι η αξία τους. Σας ευχαριστώ και αυτό με οδηγεί σε μια παρατήρηση. Όντως, από φέτος, όλες οι τραπεζικές δραστηριότητες υπόκειται στην υποχρέωση δημοσίευσης αναχώρα. Ορισμένοι φοροτεχνικοί, ο τύπος έχουν σχολιάσει τις δημοσιεύσεις μάλιστα ορισμένων τραπεζών. Εγώ πιστεύω ότι οι συγητές μας, τα μέλη που έχουν ε, συγκεκριμένες ερωτήσεις, πέρα δηλαδή από αυτές που θα μπορέσουμε να θέσουμε τώρα προφορικά, θα μπορούσαν να βασιστούν σε αυτές τις δημοσιεύσεις, ώστε ενδεχομένως να ζητήσουν διευκρινήσεις τέτοιου τύπου όπως ας πούμε το παράδειγμα των ε, ε, Παρθένων νήσων ή των ε, νήσων Καϊμάν. Εάν θέλουν διευκρινήσεις, η Κρυντία Αγρικόλ μας απάντησε ότι στην περίπτωση των Παρθένων νήσων οι θηγατρικές τις έχουν κλείσει ή κλείνουν. Για τις νήσους Καϊμάν δεν υπάρχει φορολογικό αντίκτυπος και νομίζω πως οι συνάδελφοι, εάν θέλουν να εμβαθύνουν, έχουμε εδώ τις πηγές ε, της ενημέρωσης και θα μπορούσατε να υποβάλλετε και γραπτές ερωτήσεις μετά από την ακρόαση. Και τώρα δίνω το λόγο εξ ονόματος του Άλντε στον κύριο Μίκαελ Τόιερ που είναι και συνεισηγητής. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω την κρύο Λεφέμπρο από την Γκρετία Γκρικόλ το εξή. Μία μονάδα της Κρήτη Αγκρικόλ πρόκειται ε, να πληρώσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 99,2 εκατομμύρια ε, σε πρόστιμο διότι έδωσε φορολογικές συμβουλές σε πελάτες ε, από ό,τι μάθαμε. τι έχετε να πείτε και πώς θα αποφύγετε εσείς ε, τέτοιες επιχειρηματικές δραστηριότητες ε, της Κρετά Αγκρικόλ να οδηγούν σε φοροδιαφυγή. Και θα ήθελα προς τον κύριο Χάμες από την ε, ING να ρωτήσω το εξής. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι Έχετε ε, θηγατρικές ε, σε φορολογικούς ε, παραδείσους, νήσι Κούκ, Βαρθέν νήσι, παραδείγματος χάρη. Και πώς θα εμποδίσετε εσείς να συμβάλλουν σε δραστηριότητες φοροδιαφυγής οι συμβουλές που προέρχονται από αυτά τα υποκαταστήματα. Παρακαλούμε απάντηση. Ο κύριο Λεφέμπρου. Για την ερώτηση για το αμερικανικό πρόστιμο, νομίζω ότι είναι εν η υπόθεση. Επιφυλάσσομαι για την απάντηση, αν μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα. όντω έχει δρομολογηθεί έρευνα από τις Αμερικανικές Αρχές για την χρήση ελβετικών λογαριασμών. Δεν έχω παρακολουθήσει από κοντά την υπόθεση, η οποία επαναλαμβάνει να εξελίξει και επιφυλάσσομαι. Αν μου επιτρέπετε. Πρόεδρος, είναι φορολογικό το ζήτημα ή όπως είδαμε στον τύπο την πολύκροτη υπόθεση της ε, BNP για συναλλαγές ε, με χώρες ε, που είναι στη blacklist, σε μαύρο κατάλογο από τις Αμερικανικές Αρχές ε, απάντηση. Όχι, οι Αμερικανικές Αρχές προσάπτει σε διάφορους τραπεζικούς ομίλους τη χρήση οντοτήτων, κυρίως στην Ελβετία, αν δεν απατώμε, για την απόκρυψη Αμερικανών υπηκών που έχουν φορολογική του έδρα στην, ε, στη ΣΥΠΑ. Πρόεδρος, μάλιστα θα το παρακολουθήσουμε, οπότε κατάλληλα δεν μπορείτε να μας πείτε περισσότερα αυτή τη στιγμή. CNG. Ευχαριστώ για την πρώτη σας ερώτηση. Οι εντέτητες αυτές ε, στο πλαίσιο του NG πληρώνουμε φόρους ε, στις χώρες στις οποίε δραστηριοποιούμαστε. Και πράγματι υπάρχουν κάποιες οντότητες ε, σε λεγόμενους φορολογικού παραδείσου, αλλά βρίσκονται εκεί πέρα για επιχειρηματικού όχι φορολογικού λόγους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε υποκατάστημα στο Λάβλαν. Γιατί, Γιατί έχουμε δουλειέ στην Μαλαισία και απαιτεί ο νόμος ε, να ε, έχει κάποιος υποκατάστημα στη χώρα. Οπότε για καθαρά νομικούς λόγους ε, βρισκόμαστε εκεί πέρα. Δεν χρησιμοποιείται για να μεταφέρουμε κέρδη εκεί. Για την δεύτερη ερώτησή σας, η ING και οι πελάτες της Κοιτάξτε, εμείς ε, με του πελάτες συνεργαζόμαστε, όπως είπαμε, για λόγου τραπεζικούς, όχι φορολογικού. Δεν φτιάχνουμε φορολογικά οχήματα για τους πελάτες μας. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένας επιχειρηματικό λόγος. Δεν υπάρχει κάτι το καθαρά φορολογικό. Αν δεν υπάρχει, όπως είπα, κάτι, κάποια επιχειρηματική σχέση, δεν ε, κάνουμε κάτι τέτοιο. Και το γεγονό ότι υπάρχει καμιά φορά καμία τέτοια οντότητα. Ε, για εμάς δικαιολογείται μόνο αν υπάρχει νομική απέτηση, αλλά καθαρά με κίνητρο τον ε, φόρο δεν ε, κάνουμε τέτοιες συναλλαγές. Monsieur le Directeur, euh, tout, à l'heure. είπατε προηγουμένως Ακούσαμε μάλλον τον ε, Διευθυντή της Κρετίας Αγκρικόλ να αναφέρει ότι για τον Όμιλο σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν 100 εργαζόμενοι που παρακολουθούν φορολογικές υποθέσεις και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τους ασχολείται με τις φορολογικές υποθέσεις του Ομίλου. Ε, ούτε έχουν δικαίωμα ούτε και ε, είναι η, δραστηριότητά τους να παρέχουν φορολογικές συμβουλές. Αντίθετα, ε, συγγνώμη, αντίστοιχα μπορείτε να μας πείτε για την ENG σε επίπεδο ομίλου πόσο προσωπικό έχετε που ασχολείται, είναι επιφορτισμένο με αυτές τις φορολογικές υποθέσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 20 περίπου είναι στην Ολλανδία που ασχολούνται με φορολογικές ε, συμβουλές ε, προς το κομμάτι της ENG που είναι στην Ολλανδία και ασχολούνται με το, ε, τη δομή του, του ομίλου για να συμμορφωνόμαστε με τις, απαιτήσει απαιτήσεις φορολογικής νομοθεσίας. Μετά, ανά τον κόσμο έχουμε άλλους 60 που καλύπτουν 44 χώρες. 80 το σύνολο δηλαδή, που ασχολούνται με την ε, φορολογική μας συμμόρφωση ε, σε ε, όλες αυτές τις χώρες. Άρα μας λέτε ότι είναι πάνω κάτω στο, στον ίδια τάξη μεγέθους κινείστε κι εσείς. Πολύ ωραία. Ο Φάμπιο Ντεμάζε. Äh, Ευχαριστώ. Έχω ερωτήσεις και για την Credit Agricole και για την ING και ξεκινάω με την ING ε, με την οποία συναλλάσσομαι εδώ στο Βέλγιο. Λάβαμε πληροφοριακό υλικό και εδώ πέρα γράφει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το επιχείρημα της ING ότι δεν υπάρχει φοροαποφυγή επειδή πληρώνουν φόρο εισοδήματος οι πελάτες τους ισχύει μόνο εν μέρη. Συχνά οι επενδυτές ε, σε Ολλανδία ή αλλού πληρώνουν φόρο στην πηγή με το να πηγαίνουν τα ταμεία στα Cayman Islands ε, ακριβώς ε, αποφεύγεται αυτή η φορολόγηση στην πηγή. Θα ήθελα λοιπόν μια αξιολόγηση δικιά σας αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Δεύτερον, η Κρεντή Αγκρικόλ είπε πως έχει δύο τέτοιες συμφωνίες στο Λουξεμβούργο και θα ήθελα να γνωρίζω Ε, από πότε είναι αυτές οι συμφωνίες είναι, έγιναν επί ε, Μάριος Χόλς και με ποιους εκπροσώπους της ε, Λουξεμβουργιανής κυβέρνησης ε, συμφωνήσατε. Σας ευχαριστώ. Και πάλι δύο λεπτά ο καθένας. Ε, κύριε Διευθυντά της ING, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε πελάτης μας όσον αφορά την ερώτησή σας για τα επενδυτικά ταμεία. Πράγματι, έχουμε τέτοιες δραστηριότητες. Είχαμε. Τα περισσότερα τα πουλήσαμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά να εξηγήσω την άποψή μας. Όταν προσφέρουμε επενδυτικές ευκαιρίες σε πελάτες, συχνά χρειάζεται ένα ταμείο για να διαμοιράσει τον κίνδυνο των επενδυτών. Υπάρχει λοιπόν ένας επιχειρηματικός λόγος για να παρεμβληθεί ένα ταμείο μεταξύ επενδυτών και επένδυσης. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο να διαμοιρώσουμε, όπως είπα, τον κίνδυνο. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό το φορολογικό αποτέλεσμα να είναι τέτοιο ώστε να πληρώνεται ο φόρος εκεί όπου δημιουργείται αξία. Αυτή είναι η σημαντική αρχή και το ταμείο στο οποίο αναφερθήκατε πράγματι είχε ένα τέτοιο φορολογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή οι επενδύσεις ε, φορολογήθηκαν στη χώρα όπου έγιναν και οι επενδυτές στο ταμείο φορολογήθηκαν στις χώρες όπου έμεναν αυτοί. Και το γεγονός ότι δεν υπάρχει δημιουργία πλούτου στο ταμείο το ίδιο ε, σημαίνει ότι τα, τα ταμεία θα έπρεπε να είναι φορολογικά ουδέτερα γιατί μόνο η δημιουργία αξίας θα έπρεπε να φορολογείται. Και αυτή είναι νομίζω μια αρχή η οποία ισχύει και σε άλλες ε, δομές. Μα με συγχωρείτε, λέτε πως βρίσκεται εκεί πέρα για επιχειρηματικούς λόγους αλλά δεν δημιουργεί κάποια αξία, δεν είναι κάπως αντιφατικό. Κοιτάξτε, ο, όταν λέω επιχειρηματικό στόχο, ο στόχος είναι να είναι ένα νομικό όχημα το οποίο θα συγκεντρώνει τα λεφτά. Ο διαχειριστής των κονδυλίων φορολογείται στη χώρα στην οποία βρίσκεται. Η διαχείριση των ταμείων δηλαδή γίνεται στο επίπεδο διαχειριστή των κονδυλίων, αλλά... ναι, αλλά όχι στην περίπτωση στην οποία υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας Ολλανδίας και Κέιμαν. Κοιτάξτε, ίσως είναι κάπως δύσκολο αυτό. Ε, ίσως δεν έχω καταλάβει ακριβώς εννοείται, αλλά τα περισσότερα ταμεία είναι έτσι ώστε σε τελική ανάλυση επιβάλλονται φόροι εκεί όπου δημιουργείται η αξία. Σας ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά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 Όσον αφορά ε, τις ε, ρυθμίσεις φορολογικές με το Λουξεμβούργο, σας έλεγα ότι υπάρχουν δύο φορολογικές ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί με δύο θηγατρικές μου από τη μνήμη μου. Να σας πω ότι το η πρώτη τέτοια συμφωνία υπάρχει από το 2009-2010 που έχει μπει σε κοινοπραξία αυτή η δική μας θηγατρική με μια άλλη γαλλική τράπεζα ε, και μάλλον δεν είμαι βέβαιος αλλά όντως ήταν η εποχή του κυρίου Κόλ μάλιστα και η ιδέα ήταν να πετύχουμε την φορολογική μείωση για την ε, ε, αποπληρωμή ε, του, του goodwill. Η δεύτερη η συμφωνία έχει επιτευχθεί μέσα στο πλαίσιο της διασφάλισης επιχειρήσεων που γίνονται σε δύο λουξεμβουργιανές δομές, τη δικιά μας την και μία άλλη που δεν έχει σχέση με τον όμιλό μας, έτσι ώστε η, να υπάρχει ναι, ήταν μόνο μία επιχείρηση εντός του Λουξεμβούργου που δεν πέρασε τα σύνορα και αφορούσε τον όμιλό σας, όχι τους πελάτες σας. Μάλιστα, τη δική μας ε, όμιλο και έναν εταίρο που δεν ήταν από την ομάδα μας, από τον όμιλό μας, συγγνώμη, ούτε ήταν πελάτες μας. Μάλιστα. Για τους πράσινους τώρα η κυρία Αντιπρόεδρος Εύα Ζολή. Εύα, θέλετε να θέσετε την ερώτησή σας σε καθέναν από τους ομιλητές. Μάλιστα, θα ήθελα. Θα, θα αρχίσω με τον κύριο Σίφερ της CNJ. Η πρώτη μου ερώτηση απευθύνεται σε εσά ε, από τον όμιλο ING. Έχετε θεσπίσει στις Westman Management Activities στο Λουξεμβούργο και την Ελβετία και έχετε φτιάξει και επενδυτικά ταμεία στο Λουξεμβούργο και στα νησιά Κάιμαν. Αυτά τώρα, αυτές τώρα οι δομές έχουν εξαρτητοποιηθεί και μπορούν να εγγραφούν στις χώρες όπου λειτουργούν και όπου γίνεται η διαχείριση, δηλαδή οι κάτω χώρες αυτές τις δραστηριότητες διαχείρισης επενδυτικών ταμείων τις χρησιμοποιείτε για να βοηθήσετε τους πελάτες σας να αποφύγουν ε, την φορολόγηση. Το 2013 είχατε τουλάχιστον 24 θηγατρικές στο Λουξεμβούργο. Εσείς μας λέτε ότι έχετε ε, θηγατρικές σε κάποιους φορολογικούς παραδείσους γιατί έχετε πραγματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες σε αυτές τα μέρη και ότι απασχολείται κόσμο. Μάλιστα. Αλλά γιατί χρειάζεστε 24 θηγατρικές. Σύμφωνα με τον οδηγό δίκαιης ε, οικονομίας στις κάτω χώρες, δεν δίνεται πληροφορίες όσον αφορά τα μπόνους, στη διαφάνεια και την δίκαιη φορολόγηση. Για παράδειγμα, κάποιοι από τους, ε, από τους ε, υπαλλήλους σας εξακολουθούν να λαμβάνουν ψηλά μπόνους, ε, ε, έως και 200% πάνω από το κανονικό τους μισθό εάν προωθούν επικίνδυνες συμπεριφορές. Δεν έχετε επίσης δηλώσει πολιτικής όσον αφορά την λειτουργία σας στους φορολογικούς παραδοήσους και την παροχή οικονομικών συμβουλών σε εταιρείε που είναι εγκατεστημένες στους φορολογικούς παραδείσους και δεν έχετε πολιτικές όσον αφορά τα λόμπι και τις συμπληρωμές των φόρων από τις εταιρείε. Για ποιο λόγο. Και ε, μια ερώτηση και πήρω στους δυο σας, σύντομα παρακαλώ. Μάλιστα, υπάρχουν ε, όρια στις σημερινές εκθέσεις αναχώρα και χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες να δημοσιεύονται ώστε να έχουμε πραγματικά την πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων σας. Είσαστε πρόθυμοι να αποκαλύψετε τα πλήρη ε, περιουσιακά στοιχεία κινητά και, κινητά αναχώρα και αναθυγατρική. Ποιο είναι το επενδυτικό κεφάλαιο και ποια είναι η αποτελεσματικότητα της τοπικής σας δραστηριότητας για κάθε παράρτημα. Μάλιστα, ο διευθυντής της ING. Όσον αφορά την ερώτησή σας για το Λουξεμβούργο. Το Λουξεμβούργο είναι μία από τις οικίες αγορές της ING. Έχουμε ε, δραστήριες επιχειρήσεις εκεί και απασχολούμε ένα σωρό κόσμο. Πολλές ε, συναλλαγές γίνονται καθημερινά με το Λουξεμβούργο. Το γεγονός ότι έχουμε 24 νομικές οντότητες για τόσο δραστήριες ε, επιχειρήσεις είναι κάτι το απόλυτα φυσιολογικό. Εάν δείτε το σύνολο της δομής μας έχουμε εκατοντάδες τέτοιες οντότητες, 24 για την δραστηριότητα στην οικία αγορά, δεν είναι και τόσο πολλά παραδείγματα. Επίσης καταβάλουμε το φόρο σύμφωνα με το, το, το ισχύον ποσοστό στο Λουξεμβούργο Τώρα, για τις, ε, τις εκθέσεις αναχώρα, όπως ανέφερα και προηγουμένως, υποστηρίζουμε πλήρως τις αναχώρα εκθέσεις, διότι πιστεύουμε όντως ότι αυξάνεται έτσι η διαφάνεια. Και αν δείτε την ε, ING και τις αναχώρα εκθέσεις μας, ήδη συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των στοιχείων αναχώρα. Έτσι νομίζω απήντησα στη τρίτη σας ερώτηση και σε σχέση με το ερώτημα που αφορά τις εντότητες σε φορολογικούς παραδείσους, όπως αποκαλούνται, όπως είπα και νωρίτερα, αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι να υπάρχει πάντοτε ένας επιχειρηματικός λόγος για μια συναλλαγή, αλλά και για μια δομή εντότητα. Οι φόροι συλλέγονται εκεί όπου δημιουργείται η αξία και από τη στιγμή που αυτές οι δύο σημαντικές αρχές πληρούνται, Μπορεί να υπάρχουν επιχειρηματικοί λόγοι να εργαζόμαστε με τέτοιου είδους ε, οντότητες. Αν δούμε τη σημερινή δομή της ING από εκατοντάδες νομικές οντότητες, λιγότερες από 10 απομένουν σε τέτοιες δικαιοδοσίες. Αλλά και για αυτές ακόμη, μόνο εφόσον υπάρχει επιχειρηματικός λόγος. Όπως στην Μαλαισία, που σας εξήγησα, υπάρχει ρυθμιστικός λόγος και από τη στιγμή που καταβάλλονται οι φόροι εκεί όπου δημιουργείται η αξία, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά, το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Η ερώτηση που απευθυνόταν σε εμά σε, τι αναφερόταν. Στο γεγονός ότι η έκθεση αναχώρα δεν έχει τόσο πολλές πληροφορίες, δεν είναι αρκετά ευρεία και ήθελα να σας ρωτήσω αν θα συμφωνούσατε να δημοσιεύετε και την αξία ανά επένδυση και ανά και αναχώρα. Κοιτάξτε κυρία μου, έχετε συλλογικά την ε, ρυθμιστική και νομοθετική εξουσία. Εάν μας επιβάλλεται να το κάνουμε αυτό, όπως μας επευλήθη η δήλωση των στοιχείων μας, ε, του κυκλοεργασιών μας, των κερδών μας, των φόρων μας ε, κτλ, τα δώσαμε εμείς τα στοιχεία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα λοιπόν όσον αφορά την διαφάνεια από τη στιγμή που εσείς μας το ζητάτε και το απαιτείτε. Και πιστεύω κιόλας ότι από τη, στην που θα προκύψει από την εφαρμογή που θα υποβάλει η Κομισιόν στην Επιτροπή ΜΠΕΠΣ θα το κάνουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Μάλιστα, ευχαριστώ. EFTD Μάρκο Τζάνι. Προς τους δύο ομιλητές. Ε, απευθύνομαι. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά και τις δύο, τις δύο και αναφέρεται σε μια εξήγηση για το λόγο για τον οποίο τα οχήματα ε, όσον αφορά τους τίτλους είναι σε παραδείσους φορολογικούς. Ε, στο Γκένσι για την Κρέτη Αγρικόλ και στο Ντέλαγουρ υπάρχει ένα καταπίστευμα της ING και μια ερώτηση δεύτερη για την Κρέτη Αγρικόλ. Οι μελέτες αναχώρα οι εκθέσεις αναχώρα στον ισολογισμό σας δείχνουν ότι ε, με ίδιο κύκλο εργασιών τα παραρτήματά σας στους φορολογικούς παραδείσους έχουν κέρδος 19 φορές μεγαλύτερο από αυτό που έχει που, έχουμε, που έχει ο Όμιλος στη Γαλλία. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα στοιχεία διερωτώμε πώς κάνουν οι τράπεζες για να έχουν περιθώρια παραγωγικότητα συστηματικά πιο ψηλά στους ε, που είναι εγκατεστημένα στους φορολογικούς παραδείσους σε σχέση με τον Όμιλο στη Γαλλία και από πού προέρχονται τέτοιες διαφορές όσον αφορά την απόδοση στο εσωτερικό του ίδιου ομίλου και η δεύτερη μου ερώτηση αφορά πάλι την παραγωγικότητα ανά θηγατρική. Και πάλι βλέποντας την κρεντή Αγκρικόλ, η μάλλον οι υπάλληλοι στους παραδείσους έχουν 37 φορές μεγαλύτερη αποδοτικότητα από τους υπαλλήλους στη Γαλλία. Αν δούμε τώρα τους υπαλλήλους στην Ιρλανδία και το συγκρίνουμε με τους Γάλλους, βλέπουμε ότι ο Ιρλανδός έχει παραγωγικότητα 140 φορές παραπάνω από τον Γάλλο. Αυτά τα νούμερα σημαίνουν ότι οι δεξιότητες των Ιρλανδών είναι τόσο πιο τεράστιες από αυτές των υπολείπων υπαλλήλων ή απλά αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ρυθμιστικό και φορολογικό καθεστώς ε, δεδομένου ότι η Ιρλανδία ε, παλιότερα χρησιμοποιούνταν για φοροδιαφυγή πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οι Ιρλανδοί συνάδελφοι είναι περήφανοι που είναι εκατόν τόσες φορές πιο παραγωγικοί. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση απευθυνόταν στις δύο τράπεζες, στην ING. Θέλετε να απαντήσετε στην πρώτη, παρακαλώ, εσείς. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, η πρώτη ερώτηση αφορούσε ένα ε, τράστε στο Delaware. Ναι, ποια είναι η λογική της δημιουργίας αυτού του Delaware Trust για να εκδίδει τίτλους. Ε, και να σας πω ποια είναι η λογική του Trust Delaware είναι ότι υπάρχουν νομικοί λόγοι που το χρησιμοποιούμε. Δεν οδηγεί σε μη επιθυμητό φορολογικό αποτέλεσμα. Εάν θέλ... Νομίζω εδώ πρόκειται για τίτλους ε, χρεωστικούς και εδώ έχουμε τους επενδυτές σε αυτό το μέσο και τις ε, πληρωμές σε κουπόνι για αυτούς τους ε, συμμετέχοντες. Ο εκδότης είναι η ING. Και οι αποδείξεις αυτών των κουπόνιων είναι φορολογητέα, δεν εξαιρούνται δηλαδή από τη φορολόγηση για τους επενδυτές. Τώρα, το ότι υπάρχει και το trust αυτό δεν αλλάζει κάτι. Ούτε είναι ενάντια στην αρχή ότι τα εισοδήματα θα πρέπει να φορολογούνται εκεί όπου παράγονται. Ευχαριστώ. Ο, η Κρυντή Αγκρικόλ, όσον αφορά τα, το μέσο έκδοσης του Γκέντζε, πρόκειται για το, εταιρικό, το ενοχικό δίκαιο. Δεν μπορούσαμε κάποτε να κάνουμε τέτοιου είδους ε, όχημα έκδοσης στην Γαλλία. Εάν δείτε όμως προσεκτικά, η δημοσίευση που κάνουμε στο έγγραφο αναφοράς μας λέει τα εξής σαφώς ότι το αποτέλεσμα αυτών των οχημάτων εκδοχής που βρίσκονται στο Γένζε ε, ε, λειτουργούν με εφαρμογή του γαλλικού φορολογικού δικαίου. Είναι το άρθρο 209β, καταβάλουμε το φόρμα στη Γαλλία ε, με τα, με, επί τη βάση το κύκλου των δομών στο Γκένζο. Όσον αφορά την Ιρλανδία, όπως και εσείς είδατε, είδα την έκθεση έξω την περασμένη εβδομάδα, που όντω η παραγωγικότητα σε ορισμένε χώρε συγκρίνεται. Για την Ιρλανδία απάντησα ήδη, έχουμε όντω ένα ποσοστό 12,5% φόρο ε, επί των επιχειρήσεων στην Ιρλανδία, ενώ στην Γαλλία έχουμε 38%. Ε, εκεί πρόκειται όμως για τα ταμεία ε, ασφαλιστικά, τα οποία είναι διαφανή και σημαίνει ότι φορολογούνται στην Γαλλία. Υπάρχουν όντω αποτελέσματα τα οποία δεν φορολογούνται στην Ιρλανδία σύμφωνα με τη CBCR γιατί αυτά τα αποτελέσματα φορολογούνται στην Γαλλία. Σας ευχαριστώ. Επειδή πολλοί συνάδελφοι επανήλθαν σε αυτό το σημείο, κύριε Διευθυντά, θα ήθελα γραπτός να μας στείλετε και αυτό που μόλις μας είπατε, ώστε να το κατανοήσουμε καλύτερα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε όμως τη διαφορά παραγωγικότητας ανάμεσα στη Γαλλία και την Ιρλανδία. Ευχαριστώ. Θα σας δώσω γραπτό στην απάντηση όσον αφορά αυτή την υπερπαραγωγικότητα των Ιρλανδών συναδέλφων. Είναι πολύ αγωνιστική, πολύ αγωνιστική οι Ιρλανδοί. Όσοι έχουν πάει να δουν ράγμπι γνωρίζουν πολύ καλά γιατί οι Ιρλανδοί είναι και καλύτεροι από τους Γάλλους. Ο συνάδελφος δεν είναι εδώ ο Μπράιν Χέις δυστυχώς, αλλά... Τώρα, εξ ονόματος του ΕΛΚ, ξαναδίνουμε το λόγο στην Τανούτα Χούμπνερ. Θα ήθελα Δύο σύντομα ερωτήματα να θέσω για τις ε, δημοσιεύσεις αναχώρα. Στα πλήθεια των εμπειριών σας, για τις εκθέσεις αναχώρα έχετε, εντοπίσετε ευαίσθητα ζητήματα από πλευρά εμπορικών συμφερόντων. Και δεύτερη ερώτηση, πάλι για το θέμα των εκθέσεων αναχώρα, αλλά στα πλαίσια της διευθέτησης ε, διαφορών στα φορολογικά ζητήματα. Ξέρουμε ότι η δημοσίευση πληροφοριών θεωρητικά ενδέχεται να ε, κυοφορεί το κίνδυνο επιλογής της φορολογικής βάσης σε, μια ε, χώρα όταν ε, θεωρείται ότι δεν είναι αναλογικά υψηλή η φόρη σε σχέση με την αξία που παράγεται σε αυτή τη χώρα αυτό θα μπορέσει θα μπορεί ενδεχομένω να οδηγήσει σε διαφορέ σε φορολογικά ζητήματα, διπλή φορολόγηση και ούτω καθεξή. Εσείς εντοπίζετε τέτοια ζητήματα, μήπως η βιομηχανία υπερβάλλει όταν καταγγέλει τέτοιες περιπτώσεις. Ε, ευχαριστώ, λέω πρόεδρος. Είναι η ίδια ερώτηση και προς τους δύο. Ο κύριος Μπελά, να απαντήσει πρώτος. Ναι, για τα εμπορικά συμφέροντα, αν ε, κινδυνεύουν από την υποβολή εκθέσεων αναχώρα, κοιτάξτε, δεν ε, ε, είχαμε εμεί τέτοια προβλήματα. Σε κάποιους βιομηχανικούς τομείς ενδεχομένως να είναι διαφορετική η κατάσταση, μπορώ να το καταλάβω και μπορεί. Ε, αλλά δεν, δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα την ερώτησή σας για τη διευθέτηση διαφορών. My question was that with the country by country... Για την ε, ε, έκθεση πάλι αναχώρα υπάρχει δημοσίευση των πληροφοριών και η χώρα που διαβάζει αυτές τις πληροφορίες και μπορεί να ζητάει ευρύτερη φορολογική βάση. Μήπως αυτό οδηγεί σε περισσότερες διαφορές για τη διπλή φορολόγηση. Έχετε εσείς ε, αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα για την ε, δημοσίευση των εκθέσεων αναχώρα. Εδώ και τρία χρόνια υπάρχει, εδώ και δύο χρόνια λειτουργεί πλήρως το σύστημα στην τωρινή του μορφή. Δεν αντιμετωπίσαμε τέτοια προβλήματα. Όντως, θα μπορούσαμε να ενδεχομένως να ανησυχήσουμε διότι ε, μπορεί κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες να χρησιμοποιήσουν αυτό το σύστημα Ότε, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερο, ένα μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα, ας το πω έτσι. Πρόεδρος. Αυτό είναι ταυτόχρονα ένας από τους στόχους, αλλά και ένας από τους κινδύνους ε, της μεταρρύθμισης. Τι λέει ο διευθυντής της CNG. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ως προς την, ε, ε, το θέμα της ε, δημοσίευσης ευαίσθητων πληροφοριών και τα εμπορικά συμφέροντα. Οι ε, απαιτήσει ε, της ε, CRD4 για την εκθέσει αναχώρα επιτυγχάνουν την ισορροπία ανάμεσα στην κοινοποίηση, δημοσίευση ευαίσθητων πληροφοριών και διαφάνειας. Νομίζω ότι είναι αποτελεσματική διατύπωση των διατάξεων για την εκθέσει αναχώρα. Νομίζω ότι ε, η ισορροπία παραμένει ακόμη και αν διευρυθεί το σύστημα. Από τη δική μας εμπειρία δεν έχουν δημιουργηθεί ε, διαφορές ε, λόγω αυτών των εκθέσεων. Όμως ισχύει το σύστημα μόνο από το 2014. Είναι λίγο νωρίς για να το κρίνουμε. Η αύξηση της διαφάνειας είναι κάτι θετικό, όμως θα πρέπει να έχουμε το νου μας. Ε, ε, να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στη διαφάνεια και την δημοσίευση ευαίσθητων πληροφοριών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε η Εύελιν Ρέγνερ για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Το ερώτημα απευθύνεται κυρίως στον εκπρόσωπο της Κρίντια ε, αλλά και στον άλλο κύριο και αφορά το θέμα των ενισχύσεων και των εκθέσεων ανά χώρα. Τι κάνετε όσον αφορά τις απαιτήσεις που υπάρχουν για τις κρατικές ενισχύσεις ε, όσον αφορά τις εκθέσεις αναχώρα, γιατί θα έπρεπε να αναφέρονται αυτές η Credit Agricole έχει, δεν έχει δηλώσει, με συγχωρείτε, τέτοια ενίσχυση για το έτος 2014. Το 2014 υπήρχε τέτοια ενίσχυση μορφή tax credits ή έκπτωση του κόστους ε, του μισθολογικού και γιατί δεν ε, δημοσιοποιήθηκε. Γιατί χρησιμοποιήθηκε. Μας λέτε ότι ήταν για έρευνα και ανάπτυξη. Ε, τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Αυτά. So, it's first a question to, to the... Προς την ε, Κρεντή Αγκρικόλ και μετά έχετε και άλλη με ερώτηση. Όχι, όχι, γενικά και για την, ε, προς την ΙΕΝΖΕ. Κοιτάξτε, γενικά η σχέση των εκθέσεων αναχώρα με τις ε, κρατικές ενισχύσεις. Καταλάβατε την ερώτηση, κύριε Διευθυντά. Όντως, όπως και όλες οι γαλλικές επιχειρήσεις, είχαμε tax credits Και τότε ε, δεν είχα, με θεωρήσει αυτά τα tax credits ε, ήταν επιδοτήσεις γιατί όλοι ε, είχαν, έτυχαν τις ίδιες μεταχείρισης και κοινοποίησαμε όλα τα στοιχεία. Πήραμε για την έρευνα 25 εκατομμύρια για τον όμιλο, αν θυμάμαι καλά, σε tax credit και επίσης το CICE δηλαδή είναι μείωση των εισφορών, ε, αυτό το θέσπισε η κυβέρνηση πριν από δύο χρόνια, 145 εκατομμύρια. Αυτό το tax credit είναι φορολογική ελάφρυνση για τις εισφορές ως προς τη φορολογική βάση είναι η μισθή που είναι κάτω από 3,5 ελάχιστους μισθούς, κάτι τέτοιο. Οπότε ε, μας δίνουν αυτή τη φορολογική ελάφρυνση για τις ε, εισφορές. Ως προς το, η πρώτη φορολογική ελάφρυνση για την έρευνα, ναι, κάνουμε έρευνα, μία εφαρμογή ε, της έρευνας είναι οι πιστοτικές κάρτες που έχετε όλες στην τσέπη σας. Και γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε τη φορολογική ελάφρυνση το ήλεγξε και το επανήλεγξε η φορολογική αρχή ε, ε, αυτό που κάναμε με το συγκεκριμένο κονδύλι. Ευχαριστούμε κύριο Σύπα. Πρόεδρε. Για την ING στην έκθεση του 2015 σύμφωνα με την οδηγία για τις κεφαλικές απαιτήσεις 4 ε, περιλαμβάνομαι διάφορες κρατικές ενισχύσεις γύρω στα 3, 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια ευρώ για το 2015 και το συνολικό μας φορολογικό βάρος ήταν 1,6 δισεκατομμύρια για να έχετε μια έτσι, ιδέα οπότε περιλαμβάνετε το ποσό Σας ευχαριστώ Κυρία Ρέγνερ Επιπροσθέτως, ε, ως προς την απάντηση της Κρετή Αγκρικόλ. Θέλουμε να κάνουμε τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε δύο σαφώς διακριτά ζητήματα. Έχουμε αυτό το περίφημο το σε ή ε, ε, γαλλιστή. Είναι όντως μια φορολογική ελάφρυνση, μεταφορά φόρου αν θέλετε. Δεν έχει σχέση με τον εταιρικό φορό, έχει σχέση με τις κοινωνικές εισφορές που καταβάλουν όλες οι γαλλικές επιχειρήσεις για τη χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Λοιπόν, για να ελαφρύνουμε το άχθος, ε, το βάρος ε, των ε, εργατικών, εργασιακών εισφορών για τις επιχειρήσεις, αποφάσισε η κυβέρνηση να το εφαρμόσει σε όλες τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το προσωπικό και τους μισθούς, με ένα όριο που στόχου είχε να καλύψει περισσότερο τους χαμηλούς από ότι τους υψηλούς μισθούς. Όλες οι επιχειρήσεις λοιπόν επωφελήθηκαν και δεν είναι το θέμα μας εδώ. Τώρα, για τη φορολογική ελεύθερη για την έρευνα, αντίθετα, αυτό εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητων μα. Ε, και το, η, η, λύση που βλέπω εγώ είναι το CCTV, η κοινή ενοποιημένη βάση, διότι είναι πολιτική προτεραιότητα για τα 28 κράτη-μέλη αυτό το θέμα και έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα με τον ίδιο ακριβώς ε, στόχο. Οπότε όταν ε, έρθει η στιγμή οι εισηγητές μας για το CCCTB εγώ προσωπικά θα τους πρότεινα να φροντίσουν ώστε όλοι να την χάνουν της ίδιας φυσικά προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης για την έρευνα και την καινοτομία είτε για όλους τους κλάδους είτε για Ορισμένου βιομηχανικού τομεί που ε, αναδεικνύουμε εμεί ω προτεραιότητα. Λιδού, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους και δίχως άλλη μετάβαση, όχι ότι έχουμε καθυστερήσει, αλλά θα πρέπει να διατηρήσουμε τον εντατικό αυτό ρυθμό για να μην έχουμε χρονική υπέρβαση. Ζητώ από τους εκπροσώπους της Νόρδια και της Σανταντέρ να έρθουν και να αντικαταστήσουν τον κύριο Μπαλά και Σιμπέρ που ευχαριστώ και πάλι για την συνεργασία τους. Φυσικά μπορείτε να παραμείνετε στην αίθουσα εάν το επιθυμείτε για να παρακολουθήσετε τη συνέχεια των ακροάσεων των συναδέλφων και ανταγωνιστών τους. Γίκβαλ για την Όρδεα. Καλώς ήρθατε. και η κυρία Λόπεθ Μονίθ. Μαρία. Α, Μόνικα. Μόνικα Λόπεθ Μονίθ. Η κυρία Γεκβάλη είναι εδώ. Πολύ ωραία. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ήσασταν μέσα στην αίθουσα κατά τη διάρκεια της πρώτης ακρόσης και ως εκ τούτου γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τις ακροάσεις. Προτείνω να κάνετε μία πεντάλεπτη εισαγωγική παρέμβαση. Κατόπιν θα περάσουμε σε απαντήσεις με αλφαβητική σειρά κυρία Γίκφαλ από την Νόρντεα. Πέντε λεπτά. Please. Mr. Chairman, members of the Parliament, ladies and gentlemen, thank you for the invitation αγαπητοί κύριοι Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχω σήμερα σε αυτή την ακρόαση. Ονομάζομαι Ιραντίβαλ και είμαι επικεφαλή του φορολογικού τμήματος της Νορδεά, που είναι η μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερος πάροχος χρηματοπιστωτικών ε, υπηρεσιών, ε, εταιρική τράπεζα, ε, ε, ε, τραπεζική ομίλων, αλλά και ιδιωτών. Και λειτουργούμε στις σκανδιναβικές χώρες όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, η Δανία και η Φιλανδία. Η Νόρδια απασχολεί, έχει περίπου 11 εκατομμύρια υπαλλήλους και γύρω στα 700 παραρτήματα. Η Νορτέα είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές τράπεζες με αλφα, ε, βαθμό α και είναι ανάμεσα στις 10 μεγάλες ε, τράπεζες υπηρεσιών στην Ευρώπη. Στην Νορτέα προσπαθούμε να παρέχουμε σπουδαίες ε, την εμπειρία στους, πελάτες μας με βάση ηθικές ε, προδιαγραφές που διαγράφονται στην πολιτική μας περί φορολόγησης αλλά και βιωσιμότητας όταν συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για τις φορολογικές ε, επιπτώσεις των διαφόρων προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων. Επίσης ε, φροντίζουμε ώστε να συμμορφωνόμαστε με εξωτερικές ρυθμίσεις όσον αφορά την παροχή σωστών πληροφοριών ώστε να μην παραπλανούμε τον πελάτη στην ε, διαδικασία λήψης της απόφασής του. Έχουμε μακροπρόθεσμη δέσμευση για δομημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην βιωσιμότητα. Το 2015 ξεκινήσαμε μια νέα στρατηγική βιωσιμότητα και στη διάρκεια του έτους ενισχύσαμε την νοοτροπία συμμόρφωσης και ενισχύσαμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων. Ελπίζουμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον, εμπλεκόμενοι άμεσα και δραστήρια με τις εταιρείες που χρηματοδοτούμε και τους πελάτες με τους οποίους έχουμε αγοραπολίσεις. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες για τις αποφάσεις μας τις επιχειρηματικές. Εν γέννη, καλωσορίζουμε πρωτοβουλίες που επιφέρουν σαφήνεια, συνέπεια, συνοχή, καθώς και μία γραμμίζουν τους κανόνες διεθνώς. Για της ε, πολυεθνικούς ομίλους όπως η Νορδιά, ένα συντονισμένο ε, αντιμετώπιση φορολογική είναι θετική εξέλιξη. Κατά τη γνώμη μας, άσχετα από τις πρωτοβολίες του ΟΣΑ σε σχέση με τα μέτρα για τη μετακίνηση των κερδών κτλ. Εμείς έχουμε συμβάλει δραστήρια στις διαβουλεύσεις που έγιναν. Επιπλέον συμμετέχουμε στις διαβουλεύσεις και στους γύρους διαβουλεύσεων σε σχέση με την οδηγία ε, κατά της φοροδιαφυγής της Κομισιόν καθώς και ε, συμβάλλουμε σε όλες τις συζητήσεις για εναρμόνιση. Σε, ε, συμφωνία με τις εξωτερικές μας υποχρεώσεις ε, υποβάλλουμε ετήσια έκθεση με αναχώρα αναφορά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ Κυρία μου, πιστεύω πως οι συνάδελφοι που το επιθυμούν θα σας υποβάλουν ερωτήσεις και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μόνικα Λόπεθ Μονίθ που είναι αντιπρόεδρος της Τράπεζας Σανταντέρ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας αυτή την ακρόαση. Εκτιμούμε τη δυνατότητα που μας δίνεται να είμαστε σήμερα εδώ για να συμβάλλουμε στις εργασίες αυτής της Επιτροπής. Ονομάζομαι Μόνη Καλόπεθμονής και είμαι ανώτατη ε, εκτελεστική διευθυντής και αντιπρόεδρος της από το 2015. Είμαι επικεφαλής ε, της ομάδας συμμόρφωσης και αναφέρομαι άμεσα στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Είμαι υπεύθυνη και είμαι πολύ περήφανο γι' αυτό για την προώθηση της ιδέας ε, της προσχώρησης της, ε, του ομίλου Σανταντέρ στις νομικές απαιτήσεις καθώς και στις αρχές αξίες της, του κώδικα δεοντολογίας προσαρμόζοντας συγκεκριμένε προδιαγραφές και ενημερώνοντας και πληροφορώντας τους πελάτες μας αλλά και τους υπαλλήλους μας ε, καθώς και την ευρύτερη κοινότητα. Είμαστε μια πραγματικά παγκόσμια ε, τράπεζα εγκύτητας και λειτουργούμε σε 10 γεωγραφικές περιοχές ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε 10 βασικές αγορές και έχουμε πολύ υψηλή συγκέντρωση ε, δανείων και περιουσιακών στοιχείων από τη τάξη του 60% μάλιστα. Δουλεύουμε μέσω αυτόνομων ε, θηγατρικών εταιριών που χρηματοδοτούνται δηλαδή τοπικά. Είμαστε μεγάλη αλλά απλή τράπεζα και αυτά το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας. Έχουμε λοιπόν θεσπίσει γενικές αρχές που αποτελούν την φορολογική στρατηγική της τράπεζας, της, ε, της τράπεζας Santander. Να σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, τονίζοντας κάποιες από αυτές τις αρχές. Πάντοτε πληρώνουμε την φορολογία μας ε, στο πνεύμα και στη, όχι μόνο στη διατύπωση της νομοθεσίας, υπό την αρχή ότι τα κέρδη θα πρέπει να φορολογούνται εκεί όπου γεννώνται. Εμείς ε, προσπαθούμε να εμποδίσουμε επιχειρήσεις ε, ή πρακτικές που είναι γνωστό ότι είναι προβληματικές ή που έχουν άλλους σκοπούς εκτός από την εξοικονόμηση ε, και ε, συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές και δίνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες με αληθή και πλήρη τρόπο και επιδιώκουμε τη δημιουργία μιας ε, σχέσης συνεργασίας με τις φορολογικές αρχές επί τη βάση της αρχής της διαφάνειας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Είμαστε πάρα πολύ σοβαροί όσον αφορά τη φορολογική μας ε, πολιτική και αυτό ξεκινά από το ψηλότερο επίπεδο. Το Διοικητικό μας Συμβούλιο ενέκρινε αυτή τη στρατηγική και επιβλέπει την εφαρμογή της. Έτσι έχουμε φτιάξει, έχουμε συστήσει πολύ αυστηρές διαδικασίες και ένα γενικό κώδικα διοντολογίας που καθιστά σαφές ότι δεν ανεχόμαστε πρακτικές που σημαίνει, να σημαίνουν την φοροαποφυγή εις βάρος δηλαδή της δημόσιας οικονομίας. Η διακυβέρνηση της φορολογία μας επανειλημμένω έχει βελτιωθεί με τον καιρό γιατί μαθαίνουμε από την εμπειρία μας και υιοθετούμε τις καλύτερες διεθνεί προδιαγραφές. Ω προς αυτόν έχουμε υιοθετήσει τον Ισπανικό Κώδικα Καλών Φορολογικών Πρακτικών του 2010 ε, από τους πρώτους μάλιστα. Η βασική μας αρχή φυσικά ισχύει και για τις υποχρεώσεις της φορολογικής των πελατών μας. Αυτό σημαίνει ότι στην ε, διαφήμιση αλλά και την πώληση των προϊόντων μας δεν παρέχουμε φορολογικές συμβουλές. Τα προϊόντα μας και οι υπηρεσίες μας προτείνονται και εγκρίνονται τοπικά μέσω των καταλήλων επιτροπών και σύμφωνα με τις πολιτικές του ομίλου και με την έγκριση της ε, εταιρική Επιτροπής της οποίας προεδρεύω εγώ, λαμβάνοντας υπόψη τις φορολογικές επιπτώσεις κάθε πρότασης. Επίσης εφαρμόσαμε πολιτικές αμοιβών και πρακτικές αμοιβών μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας της ρευματοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές υποχρεώσεις ε, στις διάφορες ε, χώρες. Ε, πιστεύω πως κατέστησε σαφές ότι προσπαθούμε να έχουμε μια προσεκτική επιχειρηματικά προσανατολισμένη προσέγγιση σύμφωνα με την εταιρική μας νοοτροπία απλό προσωπικό προσωπικό και δίκαιο και αυτού του είδους τις υπηρεσίες προσπαθούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας. Ε, μπορώ μόνο να σας πω ότι η Santander υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων ώστε να προληφθεί η επιθετική φορολογική πολιτική και προγραμματισμός και να προωθηθεί ισότιμο πεδίο για όλες τις επιχειρήσεις στην Ένωση καθώς και δημόσια αναχώρα έκθεση καθώς και συνεπής παγκόσμια εφαρμογή των στάνταρ του ΟΣΑ όσον αφορά την ε, διάβρωση βάσης και τη μετακίνηση των κερδών. Και βεβαίως τηρούμε το πνεύμα των συμφωνιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία που μου δώσατε να εξηγήσουμε τη θέση μας για αυτά τα σημαντικά θέματα και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ Μόνικα. Μπούρκαρτ Μπάλς είναι ο πρώτος ομιλητής εξ του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στον πρώτο γύρο θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στην εκπρόσωπο της ε, Nordea Bank. Έχω την εντύπωση πως η Nordea ε, SA έχει μητρική την Nordea Bank AB με έδρα το Λουξεμβούργο και έχει μια θηγατρική εδώ πέρα την Dentrust Management Guernsey Limited που βρίσκεται στο Guernsey. Μπορείτε να μας πείτε για ποιο σκοπό συστήθηκε αυτή η θηγατρική και τι υπηρεσίες προσφέρει στους πελάτες της. Επίσης, ε, ίσως συμφωνείτε πως η δομή αυτή η εταιρική έχει... γύρει κάποια ερωτήματα. Έχετε και ερώτηση για την Σενταντέρ. Ναι, ναι, αργότερα, αλλά θα ήθελα πρώτα να ακούσω μια απάντηση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ο λόγος για την ύπαρξη των δραστηριοτήτων μας στο Γκέντζι. Δεν ε, έχω αυτή τη στιγμή τις λεπτομέρειες πρόχειρες. Θα ήθελα να πω πως η δομή που παρέχουμε στους πελάτες μας ε, δεν ε, είναι για φορολογικούς αλλά για επιχειρηματικούς λόγους. Δεν προωθούμε κάποια φορολογικά συστήματα ή την φοροδιοφυγία αλλά ευχαρίστω να επανέλθω και να απαντήσω τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους έχουμε τη συγκεκριμένη εταιρεία, αν σας βοηθάει κάτι τέτοιο. Ωραία, ευχαριστώ. Για τους σοσιαλδημοκράτες ε, ο κύριος Κοφόντ. Α, νόμιζα ότι είχατε και άλλη ερώτηση. Μετά, μετά. Ωραία. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω και εγώ με την ε, Νορδέα. Και να ρωτήσω την κυρία Τίκμπαλ. Βλέπω πως έχετε παρουσία και στο Λουξεμβούργο μεταξύ άλλων και αναρωτιέμαι αν έχετε υπογράψει κάποιες ε, σχετικές αποφάσεις με το Λουξεμβούργο. Επίσης υπήρχε το 2015 μια περίπτωση στην οποία η Nordea Bank AB ε, εκλήθη να πληρώσει ένα εκατομμύριο, 50 εκατομμυρίων κορονών, ένα πρόστιμο, για το ότι δεν έκανε τίποτα για να προλάβει το ξέπλυμα χρήματος στην τράπεζα. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι έχετε κάνει για να μην επαναληφθεί αυτό. Και τέλος βλέπω για εσάς ότι ήσασταν διευθύντρια στην PwC στο τμήμα φορολογίας ε, από το 2004-2009 και μετά στην Ernst Young στις ε, τέσσερις μεγάλες λογιστικές εταιρείες. Κατά την άποψή σας λοιπόν μπορείτε να μας δώσετε κάποιες συστάσεις για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την διαφάνεια για όσον αφορά την φοροαποφυγή πολυεθνικών εταιρείων. Γιατί το θέμα εδώ πέρα είναι ακριβώς πώς ο τομέας, ο χρηματοπιστωτικός βοηθάει τις εταιρείες αυτές τη φοροαποφυγή. Έχετε κάποιες συμβουλές για εμάς, τι μπορούμε να κάνουμε για να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Κύριε μου, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Να ξεκινήσω με την ερώτηση για τις αποφάσεις αυτές του Λουξεμβούργου. Δεν ε, ξέρω να έχουμε κάποια τέτοια συμφωνία με τις αρχές του Λουξεμβούργου. Θα ήθελα να πω πως πληρώνουμε γύρω στο 30% φόρο πραγματικό φορολογικό συντελεστή στο Λουξεμβούργο, οπότε δεν υπάρχει κάποιο ε, επιδότηση ή φοροαπαλλαγή στο Λουξεμβούργο, από όσο γνωρίζω. Η άλλη ερώτηση ε, δεν αφορά τόσο τον φόρο, που είναι η δικιά μου η ειδικότητα και η αρμοδιότητα. Αυτό είναι πρόστιμο που μας επευλήθη για ξέπλυμα χρήματος. Έχει να κάνει με προηγούμενα έτη και τις διαδικασίες και τις ελλείψεις που είχαν. Έκτοτε έχουμε εστιάσει πολύ στις διαδικασίες αυτές και στην ενίσχυση των διαδικασιών. Οπότε θα έλεγα πως αυτά είναι εδώ και πολλά χρόνια στην κορφή της ατζέντας της διοίκησης της τράπεζας και σε όλο τον οργανισμό. Οπότε έχουμε κάνει πολλή δουλειά για να ενισχύσουμε ακριβώ αυτές τι διαδικασίε για να φροντίσουμε να συμμορφωθούμε με τους σχετικούς κανονισμού και τις διαδικασίε ε, σύμφωνα με τις οποίε πρέπει να γνωρίζουμε του πελάτε μας. Όσον αφορά τώρα την προηγούμενη μου σταδιοδρομία και τυχόν συμβουλές δεν έχω κάποιες συμβουλές. Ε, μπορώ να πω μόνο πως θεωρώ πως αυτές οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ΩΣΑ τσομπέψ ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα, πακέντα, στα πακέτα φοροαποφυγής ε, είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Αν και θεωρώ πως υπάρχει ακόμα δουλειά που μπορεί να γίνει. Αυτά, ελπίζω να απάντησα. Σας ευχαριστώ. Για, για τους ε, συντηρητικούς, ε, η Πύρκο Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μία ερώτηση προς την Νόρτεα. Και όπως και ο κύριος Κόφωτ θα ήθελα να ασχοληθώ με το ίδιο ζήτημα. Πέρσι το Μάιο σας προειδοποίησαν και 5,6 ε, εκατομμύρια ήταν το πρόστιμο, το διοικητικό πρόστιμο για την παραβίαση των κανόνων για την νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων. Η αρμόδια ε, Σουηδική Αρχή διαπίστωσε και παραθέτω τώρα σοβαρότατες ελλείψεις για την αποτροπή της δημοποίησης ε, παρανόμων εσόδων. Επίσης το 2013 για παρόμοια ε, παρόμοιες αξιόπινες πράξεις διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε συμμόρφωση με την εκείμενη νομοθεσία και γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πρώτον, γιατί ε, η Νόρντεα έχει τόσα προβλήματα για να συμμορφωθεί δηλαδή με το πλαίσιο για των κανόνων για την νομοποίηση παρανόμων εσόδων και δεύτερον. Ο Κρίστιαν Κλωσέν, ε, ανώτατος ε, αξιωματούχος στην τράπεζά σας, υψηλά βαθμό θα λέγω συγγνώμη, στην τράπεζά σας ανέφερε πως έχει αναλάβει έκτοτε η Νορδέα μέτρα για να συμμορφωθεί με αυτό το πλαίσιο. Ποια είναι αυτά τα μέτρα, και για ποιο λόγο δεν έχουν ε, ε, ως αποτέλεσμα να μην έχετε πλέον κανένα τέτοιο ρόλο και καμία δραστηριότητα που να ε, συνδέεται με την νομοποίηση ε, παρανόμων εσόδων. Ευχαριστούμε. Κυρία μου, έχετε το λόγο. Yes, thank you. Ναι, θα προσπαθήσω να απαντήσω παρότι δεν συνδέονται τα ερωτήματά σας με τα φορολογικά ζητήματα ακριβώς. Τέλος πάντων, όπως σας έλεγα, η Νορντέα ε, παίρνει στα σοβαρά φυσικά το πρόστιμο και τις ε, κατηγορίες αυτές για τις ελλείψεις. Βασιζόταν ε, οι κατηγορίες σε μια παρελθούσα περίοδο. Έκτοτε Έχουμε, δρομολογή, έχουμε θεσπίσει διάφορα μέτρα, ούτως ώστε να συμμορφωθούμε με αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχει ένα, για ολόκληρο τον όμιλο ένα πρόγραμμα στην Ορδέα για να εφαρμοστούν οι απαιτούμενες αλλαγές. Ε, δραστηριότητες κατάρτισης, ε, παραδείγματος χάρη, και ε, διάφορες διαδικασίες δέωσας επιμελίας ε, για, την, ε, για τις υπηρεσίες προς τους πελάτες. Αυτά έχω να πω. Και ελπίζω να απάντησα. Δεν μπορείτε, λέει ο Πρόεδρος, να είστε πιο συγκεκριμένοι για τις νέες διαδικασίες που δρομολογήθηκαν στην Ορντέα ώστε η παραβίαση των κανόνων περί παρανόμων εσόδων ε, να ε, είναι πιο ξεκάθαρες. Ε, αν απάντηση, ναι, μετά την τορνή ακρόαση μπορώ γραπτός να σας στείλω τα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή όχι. Ευχαριστούμε η κυρία και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής θα εκτιμήσουν δεόντως τις ε, γραπτές παρατηρήσεις. Από τους ελεύθερους νομίζω ο συνάδελφος Γκίζεκ ε, θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το ίδιο ερώτημα ήθελα και εγώ να θέσω, αλλά με προλάβανε οι συνάδελφοι. και δεν νομίζω να μας δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Προς τη Σανταντέρ και έχουμε ένα δημοσίευμα τύπου εδώ και οι πληροφορίες που λένε ότι ε, ο στόχος ήταν να κλείσουν 7 οντότητες φορολογικούς παραδείσους διατηρώντας 4 οντότητες σε περιοχές όπου υπάρχουν προγράμματα ανταλλαγής πληροφοριών με την Ισπανία. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για το τι συνέβαινε ουσιαστικά, τι συνέβη στο παρελθόν και τι προβλέπετε για το μέλλον. Απάντηση. Μάλιστα. Οι πληροφορίε είναι δημόσιες, οπότε στην ετήσια υποχρεωτική έκθεση αναφέρουμε ότι βάσει ισπανικής νομοθεσίας ο Μήλος Αντοντέρ έχει 10 θηγατρικές που ε, offshore ε, ε έδρες που όμως δεν θεωρούνται φορολογική παράδειση από τον ΩΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως πολύ σωστά είπατε, τρεις από αυτές ε, τις εκαθαρίζουμε και για τα επόμενα χρόνια ε, θα καθαρίσουμε τέσσερις. Θα έχουμε τέσσερις μόνο πλέον στο Γκέρνσε και στα, στην Ισομάν και μπορώ να σας δώσω και στοιχεία αν θέλετε. Από International Limited στο Γκέρνσε, πολύ περιορισμένη δραστηριότητα. Ε, γιατί έχουν μεταφερθεί ε, στην, άλλη εταιρεία που έχουμε στον Γκέρνσεϊ και έχουμε και άλλες δύο εταιρείε περιορισμένες ευθύνε ε, στο ΜΑΝ. Ε, οπότε με ρωτάτε γιατί δεν θα κλείσουμε στο άμεσο μέλλον και αυτές τις τρεις. Η απάντηση είναι ότι υπάρχουν νομικά κολλήματα, υπάρχουν διοικητικά ζητήματα σε σχέση με τους πρώην κατόχους ε, των θηγατρικών Μόλις διευθετηθούν ε, αυτά τα ζητήματα θα τις κλείσουμε. Το 2015 11 εκατομμύρια ευρώ ήταν το κομμάτι αυτών των οντοτήτων στο συνολικό απολυσμό. Έχουμε και πέντε υποκαταστήματα στην νησιά Κέιμενε, Μαν και Γκένσι. Ένα στο καθένα. Ε, είναι ενοποιημένοι οι λογαριασμοί στον ισολογισμό ε, των εταιριών στις οποίες ανήκουν. Δεν θεωρούνται offshore οντότητες και για τους ε, εργαζόμενους το 2015, το Δεκέμβρη, είχαμε 118 εργαζόμενους σε αυτές τις τρεις υπολοιπόμενες οντότητες. Ευχαριστούμε. Τώρα η Παλώμα Λόπεθ από την ΕΓΚΟΕ θα πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο ε, προσώπους των ε, δύο τραπεζών. Έχω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις είναι 182 ε, τα παραρτήματα των τραπεζών σας στους παραδείσους τους φορολογικούς. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μόλις δώσατε και μάλιστα έχω κάποιες αμφιβολίες για το τι ακριβώς ισχύει γιατί τα, τα, τα νησιά καημένα δεν δίνουν πληροφορίες για τις δραστηριότητε των πελατών τους. Θέλω να γνωρίζω ποιες είναι οι συμβουλές που δίνεται στις ισπανικές εταιρείες και στις εταιρείες άλλων χωρών ε, από πλευρά ε, της τράπεζάς σας για να μπορέσουν να αλλάξουν την πορεία της, ε, της νόμιμες εννοώ συμβουλές έτσι, για να αποφύγουν την μεγαλύτερη φορολογία. Θέλω όμως να επιστιάσω στην τράπεζα Τράπεζα Σανταντέρ. Στις 21 Οκτωβρίου 2015 δημοσιεύθηκε το πρόστιμο γιατί δεν έδωσε στοιχεία για ένα λογαριασμό στο πλαίσιο μιας ε, έρευνας για ξέπλυμα χρήματος. Γιατί τέτοιου είδου ε, μητρώα δεν, δεν δημοσιεύονται και γιατί δεν παρέχονται στους ε, εισαγγελείς. Δεύτερον, η διοίκηση του, του ομίλου. Έχουμε πρόβλημα όσον αφορά τα γραφεία σας ε, για, με την, ε, το σκάνδαλο που γιόλα, αλλά και τους ε, όσους πλέκονται στην υπόθεση Φαλτσάνη. Τέτοιες υποθέσεις δεν αποδεικνύουν μια πολύ συγκεκριμένη εγκύτητα με τις ισπανικές ολιγαρχίες εις βάρος της σωστής φορολογικής διακυβέρνησης και έπειτα αφορά την, δική τη δική σας διαχείριση. Στην Ισπανία το 2014 ε, ορίστηκε ψηλότερος φόρος ε, σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες. Ωστόσο, λόγω των συγκεντρωμένων απολειών της, ε, των, των αποταμιευτηρίων, των οποίων η Σανταντέρ είναι ο κύριος μέτοχος, υπήρξε μια φορο, επιπλέον φορολόγηση, ένα είδος tax ruling ανάποδο. ανάποδο. Θέλω να μου πείτε αν υπήρξε εξοικονόμηση φορολογική ή πρόκειται για στρέβλωση και μάλλον και δεν πρόκειται για στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ αυτό που κάνατε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας και θα προσπαθήσω να σας, ε, και θα σας απαντήσω στα ισπανικά στις ερωτήσεις που υποβάλατε. Η πρώτη σας ερώτηση αναφερόταν στην έκθεση Intermon Oxfam, σύμφωνα με την οποία έκθεση η Santander έχει 200 παραρτήματα σε φορολογικούς παραδείσους. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η όμιλο Santander βασίζεται στην νόμιμη, στον νόμιμο ορισμό του φορολογικού παραδείσου όπω όπως ορίζεται από το Ισπανικό κράτος, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει για την έκθεση της Oxfam. Έχουμε, όπως γνωρίζετε, έναν κατάλογο συγκεκριμένο που, ορίζεται, όπου ορίζονται η φορολογική παράδοση και έχουμε Σύμφωνα με την ε, ε, Ισπανική νομοθεσία υπάρχουν χώρες που έχουν συνάψει συγκεκριμένη συμφωνία ε, με την Ισπανία για παροχή των πληροφοριών από το 2003 και δεν θεωρούνται πλέον αυτές οι χώρες που έχουν υπογράψει τέτοιου είδους συμφωνία φορολογική παράδοση, παράδειση. Το πρόβλημα της διαφοράς των στοιχείων είναι ότι η Οξφάμα μειώνει τα κριτήρια, βασίζει μάλλον τα κριτήρια στην, στα κριτήρια ε, τα οποία χρησιμοποιεί ο οργανισμός που είναι ταυτόχρονος με τα κέρδη και δημοσιεύει μια παρόμοια έκθεση όπου υπάρχει συγκεκριμένη σύγχυση όσον αφορά τον αριθμό των παραρτημάτων που μας αποδίδει εμάς γιατί λαμβάνει υπόψη πηγές που δεν είναι ενημερωμένος. Όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή η τράπεζά μας δεν έχει καμία θυγατρική σε φορολογικό παράδειση, αν λάβουμε υπόψη τα κριτήρια του ΩΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν εφαρμόσουμε αυστηρά την Ισπανική νομοθεσία. Έχουμε παραρτήματα στο Τζέρσι, στις νήσους Καϊμάν και στο νήσο Μάν, που είναι καρπός των όσων έκανε η τράπεζα και την οργανωτική του ε, δομή. Θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνουμε υπόψη ότι η Oxfam θεωρεί φορολογικό παράδεισο και μέρη όπω το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Ουρουάη, η Ελβετία, το Πορτορίκο, η Παναμάς, η Ιρλανδία και οι Μπαχάμε που δεν θεωρούνται φορολογική παράδειση από τον ΩΣΑ. Ε, το δεύτερο ερώτημα που μου υποβάλλατε είναι η απόφαση μέσω της οποίας καταδικάζεται η τράπεζα Σανταντέρ με ένα πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ για μια υπόθεση ξεπλήματος ε, χρήματος όπου δεν έδωσε τις απαραίτητες πληροφορίες. Ωστόσο αυτό το πρόστιμο δεν έχει βάση αλλά προ το κίνητρο αυτής της ποινής προκύπτει από ελλειπή ενημέρωση όσον αφορά εμβάσματα που έγιναν σε δύο θηγατρικές της τράπεζας ε, στην Ανδαλουσία. Και το λέω αυτό γιατί τα κεφάλαια της τράπεζας είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Η κύρωση ποινή που επιβλήθηκε ήταν επειδή η τράπεζα είχε επίσης τιμωρηθεί με συγκεκριμένα πρόστιμα γιατί δεν υπήρχαν οι κατάλληλες πληροφορίες ε, μέσα στο πλαίσιο των πληροφοριών που έδωσε η θηγατρική μας. Ε, πάντως η τράπεζά μας δεν ε, έχει τιμωρηθεί για οποιοδήποτε πρόστιμο τέτοιου τύπου. Το τρίτο σας ερώτημα αφορούσε την φορολογική διακυβέρνηση και θέλω να τονίσω ότι η ευθύνη της προώθησης της φορολογικής στρατηγικής στην τράπεζα Σανταντέρ, όπως συμβαίνει σε όλες τις εταιρείες τέτοιου τύπου στην Ισπανία, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τη φορολογική στρατηγική και αναλαμβάνει την ε, υλοποίησή της. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να εντάξει και να ελέγξει όλα τους κινδύνους τους οποίους εκτίθεται η τράπεζα. Ένας εξ αυτών είναι ο φορολογικός κίνδυνος. Εδώ τελείωσε ο χρόνος σας για το τελευταίο ερώτημα που δεν μπορέσατε να απαντήσετε. Θα σας ζητήσω να απαντήσετε γραπτός. Μάλιστα. Και τώρα δίνω το λόγο εξ ονόματος των Πρασίνων στον Φιλίπ Λάμπερτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι προτιμάτε, στα γαλλικά ή στα αγγλικά, μιλώ απευθύνομαι στην κυρία του Σανταντέρ, στα ισπανικά δεν μπορώ, δεν θα μπορέσω να σας ευχαριστήσω το ίδιο είναι για μένα. Εσείς με καθησυχάζετε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, έχετε δίκιο. Ναι, πράγματι δεν λειτουργείτε σε φορολογικούς ε, παραδείσους. Ε, η Ολλανδία δεν είναι φορολογικός παράδεισος, ούτε το Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με τη λίστα του ΟΣΑ, η λίστα αυτή είναι άδεια. Δηλαδή μια εταιρεία που θέλει να πάει σε φορολογική παράδεισο δεν μπορεί να βρει. Οπότε έχω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση πόσες θηγατρικές έχετε στο Delaware που πρέπει να είναι η πιο πολυπληθής εταιρεία των ΙΠΑ έχετε. Πρώτη ερώτηση. Και η μεγαλύτερη οικονομία επίσης. Συγκεκριμένα τώρα. Έναν τρόπο που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για τη φοροδιαφυγή είναι να πουλήσουν ή να νοικιάσουν τα πλεοκής έδρα σε άλλες εταιρείες είτε σε άλλους πελάτες είτε άτομα είτε εταιρείες και βασικά χρησιμοποιώντας την ικανότητα ε, του ειδικού φορολογικού καθεστώτος τους να μπορούν ε, να πληρώνουν λιγότερους φόρους οι πελάτες τους μέσω της τράπεζας εάν, ε, από ό,τι αν ήταν οι ίδιοι δικαιούχοι. Π.χ. υπάρχουν κάποιες συμβάσεις μεταξύ ενός αγοραστή και ενός πολιτή για την διαφορά της ε, τιμής ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Υπάρχουν κάποιες ε, περιπτώσεις τέτοιων συμβάσεων όπου για τη φορολογική αρχή της ε, χώρας Α ο δικαιούχος είναι η τράπεζα, ενώ στη χώρα Β ο δικαιούχος είναι ο τελικός χρήστης. Είτε άτομο, είτε εταιρεία, είτε ίδρυμα, είτε οτιδήποτε. Και παίζοντας με τις διαφορές αυτές επιτρέπεται στον τελικό χρήστη να εποφεληθεί από τα δικά σας φορολογικά πλεονεκτήματα ως τράπεζα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω εάν η Σανταντέρ χρησιμοποιεί το καθεστώς της για να τα επεκτείνει και στους πελάτες της και τι μπορεί να γίνει για να το αποφύγουμε αυτό. Οπότε αν δεν ε, κάνετε τέτοιες δραστηριότητες, μήπως θα έπρεπε όλες οι φορολογικές αρχές να λαμβάνουν τις ίδιες ε, πληροφορίες και τι ίδιες πληροφορίε όπως οι επόπτες των τραπεζών γιατί καμιά φορά υπάρχουν λεπτές διαφορέ μεταξύ των όσων λέτε στον επόπτη σας και όσων λέτε στις φορολογικές αρχές και καλό είναι βεβαίω να λαμβάνουν όλες τις ίδιες πληροφορίε για να μην υπάρχουν αυτές οι ασυνεπίε. και μην ξεχνάτε και το όμορφο Delaware σας ευχαριστώ θα προσπαθήσω να απαντήσω είναι πολλές οι ερωτήσεις βέβαια Μια την πρώτη ερώτηση, τον Delaware δεν έχω πάει ποτέ, αλλά μου λένε πως ε, υπάρχει εκεί ένα υποκατάστημα, υποκατάστημα αλλά έχει στόχο να εκδίδει διάφορα χρεόγραφα. Και ο βασικός λόγος ε, είναι για το ότι πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται μόνο σε πολίτες των ΙΠΑ. Οπότε προτιμούν ε, κάτι στις ΗΠΑ, οπότε κάτι το οποίο έχει εκδοθεί σε ευρωπαϊκή χώρα. Γι' αυτό έχουμε το κατάστημα στον Delaware. Όσον αφορά την δεύτερη ερώτησή σας, πρέπει να πω πως ε, εμείς δεν δίνουμε φορολογικές συμβουλές ε, στους πελάτες μας. Όχι, δεν είναι ερώτηση. Είναι αν επιτρέπετε σε πελάτες σας να απολαμβάνουν τα ίδια φορολογικά προνόμια που έχει η τράπεζα. Γιατί όταν λειτουργείτε ως ε, ενδιάμεσος δεν έχετε τους ίδιους φορολογικούς κανόνες όπως ένας ε, τελικός χρήστης. Και μπορεί να χρησιμοποιείτε το φορολογικό αυτό καθεστώς για τους τελικούς σας ε, πελάτες. Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι αν χρησιμοποιείτε την τράπεζα ως φορολογικό όχημα. Ναι, ναι, αυτό προσπαθούσα να απαντήσω. Δεν δημιουργούμε κάποιες ιδιαίτερες δομές έτσι ώστε οι πελάτες μας να έχουν τέτοιες, ε, τέτοια πλεονεκτήματα. Έχουμε τη δική μας φορολογική δομή, αλλά δεν επεκτείνονται αυτά τα πλεονεκτήματα στους πελάτες μας. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα, αν θυμάστε. Υπάρχουν σχετικές δομές ε, στην ε, Ισπανία ε, για τη χρηματοδότηση πλοίων. Όλα αυτά αφορούσαν τους πελάτες. Η τράπεζα έχει μια φορολογική μεταχείριση η οποία δεν επεκτείνεται στους πελάτες. Δεν ε, πουλάμε τέτοια υπηρεσία στους πελάτες μας, ούτε θα χρησιμοποιηθεί η τράπεζα ως όχημα κάποιου πελάτη. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για το EFTT, Μάρκο Τσάνι και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση για την εκπρόσωπο της ε, Σανταντέρ. Το ερώτημά μου αφορά την περίπτωση δύο περιπτώσεις ε, φόρο αποφυγής ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο του 2015 για περίπου 100 εκατομμύρια στερλινών ε, με ένα υποκατάστημα μια θηγατρική σας στην Abbey National Treasury Services και πρόκειται για ένα λάθος υπολογισμό των ε, swaps ε, τα οποία καταγράφηκαν ως απώλειες οι οποίες άρα θα είχαν κάποια έκπτωση φόρου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν εάν η τράπεζα χρησιμοποιεί, χρησιμοποίησε στο παρελθόν τέτοια συστήματα έκπτωσης ε, των ε, ζημιών που είχε σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Και το δεύτερο ερώτημα αφορά την ε, Banco Santander Brazil SA που έχει έδρα στο Grand Cayman. Είναι ένα όχημα που χρησιμοποιεί συνήθως η Santander για εκδόσεις κάποιων χρεογράφων και γνωρίζουμε πως αυτές οι εταιρείες ε, στα Κέιμαν έχουν μία περίοδο φόρο 20 με 30 ετών. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μας διαφωτίσετε για την εταιρεία αυτή, το όχημα αυτό, το εταιρικό στα νησιά Κέιμαν. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Για την πρώτη ερώτηση αναφερθήκατε στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν κάποιες ε, συναλλαγές ε, ιστορικές της Abbey National, την οποία αγόρασε η Santander και έγιναν πριν ε, η Santander UK συνυπογράψει τον κώδικα φορολογικών πρακτικών το 2010. Ήταν νόμιμες λοιπόν οι συναλλαγές όταν έγιναν και απλά αντικατόπτριζαν κάποιες λογιστικές πράξεις ε, που όπως είπα όταν έγιναν ήταν νόμιμες. Οπότε υπήρχαν κάποιες τεχνικές πτυχές και θέλαμε ακριβώς να έχουμε την βεβαιότητα για το εάν ε, ε, ήταν ε, σύνομες. Οι συζητήσεις αυτές λοιπόν είναι από το 2010 και προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιες ε, λύσεις με τις φορολογικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2015 είχαμε μια αρνητική απάντηση και αποφασίσαμε να μην προσβάλλουμε την απόφαση των αρχών. Για το δεύτερο ερώτημα σας είπα ήδη πως έχουμε υποκατάστημα στις ε, νήσους ε, Κέιμαν της ε, Σανταντέρ Brazil αλλά δεν χρησιμοποιείται για παροχή υπηρεσιών στους πελάτες χρησιμοποιείται μόνο για λόγους hedging για τις συναλλαγματικές συναλλαγές του βραζιλιανικού ρεάλ με το δολάριο Μάλιστα. Για... Όσον αφορά τα νήσου Καϊμά, να σα θυμίσω ότι στην πρώτη πρόσκληση που είχαμε αποστείλει είχαμε μια αρνητική απάντηση από πλευρά των αρχών. Δεν μπορούσαν να είναι παρόντες εκπρόσωποι των νήσων αυτών ε, και όπως ε, σας είπα έκανα μια δεύτερη έκανα μια δεύτερη πρόσκληση και θα ήταν ενδιαφέρον να θέσουμε άμεσα στου ηθήνοντες τον Ίσον Καϊμάν τις ερωτήσεις αυτές που έλαβαν μερικές απαντήσεις μόνο απόψε. Και τώρα δίνω το λόγο εξ του ΕΛΚ στον κύριο Μπάλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να απευθύνομαι τώρα στην εκπρόσωπο της Σανταντέρ. Δύο ερωτήσεις έχω. Πρώτον, για το θέμα του ξεπλήματος χρήματος. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο ποιες προδιαγραφές ακολουθεί η Σανταντέρ για τις διαδικασίες εντός της ε, τράπεζας, ειδικά όσον αφορά τις δραστηριότητε σας στη Λατινική Αμερική. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πώς είναι οργανωμένες σχετικές αναφορέ και στα κεντρικά σα στην Ισπανία. Δεύτερη ερώτηση. Είπατε πως δεν ε, έχετε κάποιες φορολογικές δομές και δεν ε, δίνετε φορολογικές συμβουλές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια προϊόν δημιουργείται. Μπορεί κανείς να πει πως ε, εντάξει δεν κάνετε φορολογικές ε, συμβουλές αλλά από την άλλη πουλάμε κάποια προϊόντα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι κάνετε και ποια νέα προϊόντα σχεδιάζετε και χρησιμοποιείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σε σχέση με την πρώτη ερώτηση για τις διαδικασίες EML. Έχουμε ένα ε, ε, εταιρικό πλαίσιο κατά του ξεπλήματος χρήματος ε, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες μας τις θεγατρικές και κάθε διοικητικό συμβούλιο στις διάφορες χώρες όπου λειτουργούμε πρέπει να τηρούν αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο. Χρησιμοποιούμε το ίδιο είδος τεχνολογίας για του στόχου AML σε όλες μας τις ε, ε, εταιρείε, ε, πράγμα που μας βοηθά να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και πρακτικές ανάπτυξης στις διάφορες ομάδες. Αν και οι βασικές απαιτήσει όσον αφορά την ταυτοποίηση του πελάτη, την τμηματοποίηση των πελατών, ανάλογα με τον κίνδυνο γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Ε, για, δικά για τους πελάτες μας στην Λατινική Αμερική θα πρέπει να σας πω ότι είναι οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν είτε είναι offshore είτε είναι, offshore, είτε είναι onshore για την ιδιωτική τραπεζική. Το ίδιο ισχύει για έναν πελάτη στο Μαϊάμι όπως ισχύει και στην Ισπανία. Για έναν πελάτη στην Ισπανία. Τώρα, Όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, όταν σχεδιάζουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που θα πουλήσουμε στους πελάτες, ποτέ δεν λαμβάνουμε υπόψη το στοιχείο του φόρου ως ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έχουμε μια επιτροπή, της οποίας εγώ προεδρεύω, όπως σας είπα, όπου αξιολογούμε και επικυρώνουμε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία προσφέρεται στις χώρες όπου ε, λειτουργούμε. Όλα αυτά τα προϊόντα δηλαδή, άσχετα με το αν θα πουληθούν στη Βραζιλία, στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία, Πορτογαλία πρέπει να επικυρωθούν από την Επιτροπή. Όλες οι, όλοι οι τομεί που έχουν λόγο για το λόγο προϊόν είναι μέλη της Επιτροπής, πρέπει να δώσουν τη γνώμη τους. Έχουμε δηλαδή εκπρόσωπο για τους φόρους, αλλά έχουμε το νομικό, το εκπρόσωπο της νομικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας ε, αρμόδιας για το κίνδυνο και ούτω καθεξής και όλοι πρέπει να γνωμοδοτήσουν. Εξασφαλίζουμε βέβαια το σωστό σχεδιασμό και τη σωστή εξήγηση στους πελάτες μας σε σχέση με την φορολόγησή του. Αλλά δεν σχεδιάζουμε ένα προϊόν μόνο και μόνο επειδή δίνει φορολογικό πλεονέκτημα στους πελάτες. Σας ευχαριστώ. Τέλος, από την, ε, τους σοσιαλιστές. Καλησπέρα σας. Εγώ θέλω να απευθυνθώ στις δύο κυρίες που αντιπροσωπεύουν αυτές τις δύο τράπεζες. Καταρχάς να τους παρουσιάσω μια πολιτική, ένα πολιτικό προβληματισμό και μετά δύο τεχνικές ερωτήσεις. Ο πολιτικός προβληματισμός είναι ότι όπως γνωρίζετε εδώ βρισκόμαστε γιατί ολόκληρη Ευρώπη υποφέρει από κοινωνική ανατραχή λόγω της φοροδιαφυγής των μεγάλων εταιριών, της ψηφιακής οικονομίας κτλ. Αλλά είναι αλήθεια ότι οι τράπεζες ε, είναι μέσα σε αυτή την απαξίωση την κοινωνική που είναι πολύ μεγάλη μετά από την οικονομική κρίση που περάσαμε. Δηλαδή ο κόσμος είναι εκνευρισμένος κατά των όσων φοροδιαφεύγουν και κατά των τραπεζών γιατί επιπλέον εκείνες ε, για τον κόσμο φέρουν ε, μεγάλη ευθύνη και πέρα από το ρόλο που έπαιξαν ε, όσον αφορά την, το ξέσπασμα της κρίσης. Αυτό μας οδηγεί εδώ. Θα ήθελα να γνωρίζω αν το έχετε συνειδητοποιήσει ότι όλες, αυτές, όλες οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές οντότητες για να λειτουργήσει η οικονομία και η αγορά είναι αυτές που θα πρέπει να δώσουν το καλό παράδειγμα για τη διαφάνεια και τη συνεργασία την φορολογική που μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί αυτό. Ε, και έτσι οδηγούμε στα ερωτήματά μου. Όταν κάποιος από τα, κάποιο από τα παραρτήματά σας, τις ιατρικές σας, ε, οπουδήποτε και αν λειτουργεί, Έρχονται άνθρωποι που δεν είναι υπηκόοι αυτής της χώρας και ανοίγουν έναν λογαριασμό, ένα τρέχοντα λογαριασμό ή ένα συλλογικό λογαριασμό που επενδύει. Ποια είναι η συνεργασία με την εταιρεία αυτή των μη υπηκόων, των αλλοδαπών. Τι κάνετε εσείς λοιπόν με τις εταιρείε τις εθνικές των ανθρώπων που άνοιξαν λογαριασμού, με τις χώρες ε, ε, στις από τις οποίες προέρχονται. Ε, και, δε, και η άλλη μου ερώτηση έχει να κάνει με κάτι που συζητά το Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό. Είναι πιθανό τον επόμενο χρόνο στην Ευρώπη να υπάρχει ένα είδος νομοθεσίας και επιβάρυνσης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αυτοί οι χώροι, οι αδιαφανείς, οι offshore, θα είναι ο χώρος από όπου θα λειτουργείτε για να αποφύγετε αυτήν την επιβάρυνση. Εκεί όπου δηλαδή οι ευρωπαϊκές χώρες θα το επιβάλλουν. Θα, τι θα κάνετε, θα οδηγηθείτε σε νέα αύξηση των αδιαφανών φορολογικών χώρων. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Κίκβαλ για να αλλάξουμε λίγο. Δύο λεπτά έχετε. Ευχαριστώ. Για το πρώτο σας ερώτημα, νομίζω ότι το ξαναθήξαμε αυτό το ερώτημα, διότι έχουμε τη διαδικασία που ισχύει για ολόκληρο τον όμιλο, ανεξαρτήτως προέλευσης του ε, πελάτη, του το προέλευσης του πελάτη. Έδωσα την απάντηση, νομίζω. και υπάρχει υποχρέωση για τον πελάτη να ε, συμμορφούνται με την φορολογική νομοθεσία και να υποβάλουν τα στοιχεία του στις φορολογικές αρχές κάθε χώρα. Σε σχέση με τη δεύτερη ερώτησή σας μπορείτε να την επαναλάβετε ναι, η δημιουργία μιας επιβάρυνσης προλογικής στις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ε, θα οδηγήσει στις τράπεζες όταν λειτουργούν στις, στα χρηματιστήρια στις χρηματιστηριακές αγορές. Αυτό θα οδηγήσει στην αύξηση των αδιαφανών φορολογικών χώρων στα offshore. Αύξηση των offshore ή όχι. Μάλιστα. Για τον φόρο επιχρηματοπιστωτικών συναλλαγών Διότι σε, διαβούλε... Ε, σε γύρους διαβούλευσης νομίζω ότι το έχουμε ξαναπεί αυτά. Νομίζω ότι μιλάμε για, μια, για ένα εφάπαξ, για έναν μάλλον ενιαίο συντελεστή για ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά δεν έχω προβλέψει σε σχέση με το μέλλον. Madame. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με τον πρώτο σας προβληματισμό θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα και οι τράπεζες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα καλόφημοι από κοινωνική άποψη. Δεν είναι εύκολο το θέμα, αλλά εργαζόμαστε για να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε αυτή την κοινωνική ε, αξιοπιστία που δυστυχώς στη διάρκεια των ετών της κρίσης έχουμε χάσει. Ένα θέμα το οποίο εμείς στηρίζουμε στην Τράπεζα Σανταντέρ είναι η ανταλλαγή των πληροφοριών και σε αυτή τη γραμμή οι νομοθεσίες όπως η ΦΑΤΚΑ ή η CRS ε, μας βοηθούν ε, όντως στο να θεσπιστεί ανταλλαγή πληροφοριών όχι μόνο εντός της Ένωσης αλλά και σε διεθνές επίπεδο και όντως ε, οι τράπεζες που λειτουργούν σε πάρα πολλές χώρες και η δική μας τράπεζα υιοθέτησε μάλιστα πρώιμα αυτήν την νομοθεσία νομοθεσία έτσι ώστε να λειτουργήσει και για τις λατινοαμερικανικές ε, χώρες. Επιπλέον ε, μας βοηθά αυτό να ε, προωθήσουμε τις πληροφορίες και στα τοπικά παραρτήματα και αυτό μας δίνει την εγγύηση πως οι πελάτες μας πληρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Τώρα, όσον αφορά τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ε, εμείς ήδη, για μας ήδη ισχύει σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χώρο που να μετακινήσουμε τις δραστηριότητες μας. Το είπαμε από την αρχή, είμαστε μια τράπεζα εγκύτητας ε, ε, και τώρα α πούμε στην Πολωνία θα επιβληθεί αυτή η φορολογία, το πάθαμε και στην Ισπανία με την ε, φορολόγηση των καταθέσεων ε, ε, θα θέλαμε ε, οι κρατικές επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη ότι δεν είναι οι τράπεζες μόνο που οφείλουν να συμβάλλουν στη δημόσια οικονομία, αλλά όλοι θα έπρεπε να συμβάλλουν το ίδιο. Πάντως δεν έχουμε προγραμματίσει να μετακινήσουμε τις δραστηριότητε μας κάπου αλλού, γιατί όπως σας είπα η παρουσία μας offshore είναι πολύ περιορισμένα και θέλουμε μάλιστα να περιορίσουμε, να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο περισσότερο τα παρατήματά μας offshore. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε. τις ερωτήσεις ε, για το δεύτερο πάνελ ε, και ε, σας ευχαριστούμε κυρίες μου για τις απαντήσεις. Ε, περιμένουμε δε γραπτά ή πρόσθετα στοιχεία, κυρίως από πλευράς Νορδεα. ποιες διαδικασίες ε, θέσπισε ε, ο όμιλός μετά από τις εντοπιστήσεις ανομαλίες σε σχέση με την καταπολέμηση του, του, της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων. Ερωτήκατε πολλές φορές για αυτό το ζήτημα. Ακριβώς τι περιέχουν αυτά τα μέτρα και Επίσης δεν απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις κυρία Παλώμα Λόπες για την ε, απόφαση για σας και άλλες επιχειρήσεις σε σχέση με την ε, μείωση του φόρου επί των κερδών. Ε, σχάτως. Ιδού, σας ευχαριστώ και σας προτείνω να κλείσουμε και αυτό το δεύτερο πάνελ. Κυρίες μου, σας ευχαριστώ και όπως είπα και ε, στους υπόλοιπους συναδέλφους μπορείτε να παραμείνετε στην αίθουσα. Και τώρα, UPS και Unicredit ακολουθούν. Ο κύριος Πινιό, εκτελεστικός διευθυντής και διευθυντής ε, της εφορολογικής υπηρεσίας ε, UBS, είστε ε, μέσα στην αίθουσα και ο κύριος Τσεκάτσι και ο υπεύθυνο για τα φορολογικά ζητήματα της Unicredit.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 Ναι, ήσασταν ε, στις ε, ε, υπόλοιπες ακροάσεις παρόντες και καταλάβατε τους κανόνες βάσει των οποίων διοργανώνουμε αυτές τις ακροάσεις γιατί επιλέξαμε τα δικά σας πιστοτικά ιδρύματα. Πήραμε, επιλέξαμε τα σημαντικότερα ιδρύματα της Ευρώπης για, με τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί και μία ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Και... Έχουμε μια πεντάλεπτη εισαγωγική παρουσίαση αρχικά. Παρουσιάζεται εκεί πέρα την ε, πολιτική φορολογικού σχεδιασμού του ομίλου σας και τις συμβουλές ενδεχομένως που παρέχετε στους πελάτες σας για φορολογικά ζητήματα και κατόπιν θα σας δηθεί να απαντήσετε σε ερωτήσεις ε, όλων των μελών της Επιτροπής μας που εκπροσωπούν διάφορες πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Πινιό, UBS. Κύριε Διευθυντά, τον λόγο.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 σας ε, ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα στη UPS να έρθει σήμερα και να συμμετάσχει στις εργασίες Επιτροπής για αυτό τόσο σημαντικό ζήτημα. Η UPS είναι παγκόσμια τράπεζα, η έδρα είναι στην Ελβετία και η στρατηγική της είναι η διαχείριση στοιχείων, ε, περιουσιακών στοιχείων και ε, έχουμε φυσικά και άλλα υποκαταστήματα που είναι, δραστηριοποιούνται στην επενδυτική στρατηγική. Ποια είναι η επιχειρησιακή μας στρατηγική βοήθεια βοηθούμε ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ως ένας υγιής χώρος ε, συναλλαγών ε, για να τονωθεί η ανάπτυξη ε, και το ευσύν μέσα από τις δραστηριότητες του ομίλου μας. Και επίσης ως προς τις δραστηριότητες μας Έχουμε σε περισσότερα από 40 υποκαταστήματα σε 12 χώρε και 10.500 συνεργάτε. Προσφέρουμε πολύτιμε υπηρεσίε στου Ευρωπαίου καταναλωτέ. Δεν δημοσιεύουμε συγκεκριμένε πληροφορίε. Μπορώ να σα πω όμω ότι ε, η περιοχή στην οποία εντάσσεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί στο 22% του συνολικού μα εισοδήματο για το 2015. Οπότε είναι υψή τη σημασία αυτά που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον όμιλό μα Από παρελθούς εμπειρίες ε, διαπιστώνουμε ότι η διαφάνεια και απόλυτη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία είναι βασικά στοιχεία ώστε να επικρατεί ένα θετικό επιχειρηματικό πνεύμα και να δημιουργείται προσθέμενη αξία για τους μετόχους καταναλωτές και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκομένους φορείς. Παρότι ακόμη είμαστε στη διαδικασία διερεύνης και διευθέτησης φορολογικών ζητημάτων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάνει ε, σημαντικά συγκεκριμένα και αποφασιστικά βήματα ώστε να συμμορφωθούμε με όλες υποχρεώσεις έχουμε ως προς τους εμπλεκόμενους φορείς ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε εσωτερικό κώδικα ε, δεοντολογίας που μπορείτε να συμβουλευτείτε στην ιστοσελίδα μας και η UPS δεν εξετάζει μόνο πότε είναι νόμιμο κάτι αλλά και πότε κάτι είναι ηθικό καταβάλουμε το φόρο που μας αναλογεί σε όλες τις ε, δικαιοδοτικές επικράτησεις όπου δραστηριοποιούμαστε και οι πελάτες μας ε, δεν φοροδιαφεύγουν ε, και υποβάλλουν όλα τα πετούμενα στοιχεία. Δεν συμμετέχουμε σε εμπορικές συναλλαγές όπου ξέρουμε ότι οι φορολογικές συμφωνίες οδηγούν σε απόκρυψη πολύ σημαντικών στοιχείων. Έχουμε ένα εσωτερικό κώδικα φορολογικής διοντολογίας, εκείνο το πλαίσιο που καθοδηγεί τις αποφάσεις μας Έχουμε πέντε βασικές αρχές μας σε αυτό τον κώδικα. Πρώτον, συμμορφούμαστε πλήρως με τις βασικές αρχές χωρίς καμία εξαίρεση. Δεύτερον, ε, διευθετούμε τις φορολογικές μας υποθέσεις ώστε να έχουμε ε, βιώσιμη προσθέμενη αξία για τον καταναλωτή. Τρίτον, θα επικρατεί η διαφάνεια και άμεση επικοινωνία, κοινοποίηση στοιχείων με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Τέταρτον, δεν θα εμπλακούμε σε δραστηριότητες και προϊόντα που δεν έχουν εμπορικό σκοπό τρόπο και πέμπτον όλες οι δραστηριότητες θα ελέγχονται σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, μεταγενέστερα για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με αυτόν τον κώδικα δεοντολογίας. Έτσι διαχειριζόμαστε τις δραστηριότητες ε, της UPS ε και των πελατών μας. Κάνουμε λεπτομερή αναθεώρηση όλων των ε, στοιχείων που σχετίζονται με τις συναλλαγές σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας. Χρησιμοποιούμε εξωτερικούς συμβούλους, ούτως ώστε να κατανοούμε πλήρως την εφαρμοστέα νομοθεσία και έτσι λαμβάνεται η απόφαση αν γίνεται, αν δίνεται η έγκριση έγκριση για μια δραστηριότητα και ε, ε, ε, αυτή η έγκριση προέρχεται από μένα ή από τους προϊσταμένους μου ανάλογα με την περίπτωση. Ε, φορολογικές θέσεις ε, ε, εγκρίνονται μόνο όταν έχουν υψηλό ποσοστό επιτυχίας και όλα αυτά γίνονται σε απόλυτη διαφάνεια. Επίσης, τακτική διαβούλευση με φορολογικές αρχές, τους ώστε να εφαρμόσει σωστά η εφαρμοστή νομοθεσία και να έχουμε τα πετούμενα στοιχεία για να λάβουμε τις αποφάσεις μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της UPS συμμορφώνεται απολύτως με αυτές τις πέντε αρχές και υπάρχει απόλυτη λογοδοσία σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Θεωρούμε ότι οι φόροι είναι το τίμημα κάθε πολιτισμένης κοινωνίας ε, και ε, είναι ακρογωνιώ λίθο ε, της σωστού εταιρικού γίγνεσθε, αν θέλετε, το να υπάρχει αυτό το ήθο και να αντιτηρούμε αυτού του κανόνες. Ευχαριστούμε κύριο Τσεκάτση. Mr. Chairman, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ που μας καλέσατε και για την ευκαιρία που μας δίνεται να έρθουμε σήμερα σε επαφή με τους Ευρωπαίους νομοθέτες και να περιγράψουμε το πόσο ανταποκρινόμαστε στις φορολογικές μας υποχρεώσεις. Ήθελα να περιγράψω λίγο τον όμιλο Unicredit. Η Unicredit έχει ρίζες 17 ε, χώρες, προφανώς είναι και σε άλλες έχει πάνω από 125.000 υπαλλήλους, πάνω από 32 εκατομμύρια πελάτες στην Ευρώπη και είναι μία από τις 30 παγκόσμιες συστημικές τράπεζες. Γι' αυτό έχει για μας μεγάλη σημασία για να μπορούμε να δραστηριοποιούμαστε με ένα επίπεδο νομικής βεβαιότητας για την φορολογία και παρά το ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι περίπλοκο και βέβαιο, να αντιμετωπίζουμε σωστά τις φορολογικές μας υποχρεώσεις. Πέρα από όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες και πόρους που υπάρχουν για να συμμορφωνόμαστε με τα φορολογικά, έχουμε εταιρική ευθύνη σε όλα μας τα επίπεδα όσον αφορά τον φορολογικό κείμενο. Υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφοράς που περιλαμβάνει πολύ σημαντικές δεσμεύσεις. Να σας τις αναφέρω οι υπάλληλοι δεν πρέπει να πολλούν ή να προσφέρουν γραπτός ή προφορικός επενδυτικά προϊόντα ή άλλα προϊόντα ε, μόνο και μόνο επειδή ωφελούν φορολογικά τον πελάτη ή άλλους αντισυμβαλωμένους. Ο Όμιλος δεν πρέπει να κάνει συναλλαγές ε, με στόχο την ε, φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή οι δραστηριότητες του ομίλου πρέπει να υποστηρίζονται από έναν πραγματικό επιχειρηματικό σκοπό και μια συναλλαγή που έχει στόχο την παράκαμψη των φορολογικών διατάξεων ή την ανάκτηση φόρων απαγορεύεται. Οι πληροφορίες που δίδονται στις φορολογικές αρχές και άλλους αρμοδίους φορείς πρέπει να είναι πλήρης και αληθής. Απαγορεύεται να παρεμποδίζονται οι δραστηριότητες των αρχών αυτών κατά τη διάρκεια των φορολογικών ελέγχων και επιθεωρήσεων. Επιπλέον, προσφάτως ε, καταλήξαμε σε μια παγκόσμια πολιτική ένα φορολογικό πλαίσιο και έτσι καθορίζεται η φορολογική πολιτική της κάθε νομικής προσωπικότητας του ομίλου και καθορίζεται ποιος ο ρόλος της κάθε εταιρεία εντός του ομίλου σύμφωνα με τα όσα μας λέει ο ΩΣΑ. Και είναι υποχρεωτική η σύσταση ενός πλαισίου φορολογικού έλεγχου. Πρακτικά όμως πώς συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες τους εσωτερικούς το 2010 ξεκινήσαμε υπογράφοντας εθελοντικά τον κώδικα πρακτικής για την φορολογία των τραπεζών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2014 μόλις η Τράπεζα της Ιταλίας έβγαλε τους δικούς της ε, κανόνες. Επίσης ε, ακολουθώντας τα πρότυπα του ΩΣΑ, η Unicredit άρχισε να επενδύει για να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο διαχείρισης φορολογικού κινδύνου. Αυτό σημαίνει πως και ως φορολογούμενοι και ως ενδιάμεση έχουμε κάποιες πολιτικές ε, συμμόρφωσεις. Οπότε έχουμε μια παγκόσμια πολιτική για να συμμορφωνόμαστε και με το γράμμα και με το πνεύμα της νομοθεσίας σε όλες τις χώρες αλλά επίσης εφαρμόζουμε εκθέσεις αναχώρα παγκοσμίω και έχουμε μια στιβαρή πολιτική για τις δικαιοδοσίες εκείνες που δεν συνεργάζονται και έτσι σε κεντρικό επίπεδο ή αναχώρα εξετάζουμε κάθε συναλλαγή που περιλαμβάνει τέτοιες δικαιοδοσίες. Επίσης είδαμε το ζήτημα των νέων προϊόντων στο πλαίσιο αυτό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε κύριε Διευθύντα. Τον λόγο τώρα οι βουλευτές και για το ΕΛΚ πρώτα ο Μπουρκχάρτ Μπάλτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και την προηγούμενη φορά θα απευθύνω μια ερώτηση στον εκπρόσωπο της ε, UBS και μετά στον εκπρόσωπο της UniCredit για την UBS. Από πέρσι όλες οι τράπεζες υποχρεούνται να δίνουν εκθέσεις αναχώρα. Κάποιες άλλες τράπεζες δεν εδώ και πολύ καιρό και βεβαίως ε, αυτά δεν δημοσιοποιούνται αλλά πηγαίνουν εμπιστευτικά στην Κομισιόν οπότε ήδη έχετε εμπειρίες ε, σχετικές θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω σήμερα. Ε, για το 2014 βλέπουμε δεδομένα για δραστηριότητε σε 14 ε, χώρες, όμως όχι για την Ελβετία, όχι για τη ΣΥΠΑ, το Χονγκ Κόνγκ και κυρίως δεν βλέπουμε κάτι για τη Σιγκαπούρη. Ποιε είναι οι εμπειρίε σα με τις εκθέσεις αναχώρα και κυρίως πόσο πλήρης είναι η εικόνα όταν ε, δεν βλέπουμε τη δραστηριότητά σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά όταν μιλάμε για τη μετατόπιση δραστηριοτήτων ε, στην Ασία, ανέφερα ήδη τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κόνγκ. Ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά. No, thank you. Uh, UBS has been subject to CRD4 reporting. Το UBS τηρεί για τις ρυθμισμένες οντότητες από το 2014 όλες τις απαιτήσεις της CRD4. Και δεν υπάρχει ε, κάτι αντίστοιχο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με το CRT4. Ε, από το 2016 όμως που άρχισαν να αρχίσουν οι κανόνες για τις εκθέσεις αναχώρα, θα αλλάξει η κατάσταση για μια ελβετική τράπεζα σε παγκόσμιο επίπεδο και θα συμμορφωθούμε πλήρως με αυτούς τους κανόνες. Εμείς δεν έχουμε μετατόπιση βάσης σε καμία περίπτωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Βασιζόμαστε σε οικονομική πραγματικότητα. Δηλαδή, οι οικονομικές μας δραστηριότητες με φυσιολογικό τρόπο παράγονται εκεί όπου έχουμε εργαζομένους και ε, είναι σε αγορές ε, και σε καμία περίπτωση δεν έχουμε θηρίδες ε, και εικονικές εταιρείες κτλ. Για το 2017 όταν θα δημοσιεύσουμε τις εκθέσεις για το 2016 οι φορολογικές αρχές θα μπορέσουν με απόλυτη διαφάνεια να δουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται από πλευρά CBCR. Απαντώ κύριε Μπούλς στην ερώτησή σας, επερώτηση. Μια ερώτηση ακόμα. Σωστά είπατε πως δεν υπάρχει νομική υποχρέωση. Μπορούμε να αναμένουμε στο προσεχές ε, μέλλον παρόλα αυτά να μας δώσετε τέτοια στοιχεία για τις αγορές ε, κλειδιά της ε, τράπεζάς σας. Νομίζω πως κάτι τέτοιο θα ήταν ενδιαφέρον. Κύριε Διευθυντά. Generally speaking, uh... ε, γενικά, ε, ξαναλέω, οι κανόνες BRC ε, ε, είναι εφαρμόστε και ούτως ή άλλως σε εθελούσια βάση ε, εξετάζουμε τη δυνατότητα να δημοσιεύουμε πληροφορίες για όλα τα υποκαταστήματα και τις ε, παγκοσμίως. παγκοσμίω. Σε σχέση τώρα με την δημοσίευση των πληροφοριών, αυτό σκεφτόμαστε όπως και οι υπόλοιπε επιχειρήσεις, όχι μόνο για την Αμερική αλλά και για τον κόσμο. Εξετάζουμε λοιπόν ε, να δούμε εάν, ε, ποιο, ποιο είδους πληροφορίες μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους ανταγωνιστές μας. Δεν νομίζουμε ότι συμβαίνει αυτό, αλλά αποτιμούμε τώρα τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Ξαναλέω, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε εθελούσια βάση, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να υποβάλουμε εκθέσεις ανά χώρα. Όχι ότι υπάρχει νομική απέτηση, αλλά δεν θέλουμε να είμαστε και οι πρώτοι που θα το κάνουμε. Εάν γίνει κοινό τόπο και, ε, ε, ε, και πρακτική, θα ακολουθήσουμε κι εμείς. Πρόεδρος, υπάρχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του να είναι κάποιος πρώτος σε σχέση με τη φήμη του. Από τους σοσιαλιστές η Ευελίνα Ρέγνα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα μια ερώτηση στον εκπρόσωπο της UBS και μετά μια και στους δύο. Στα ΜΜΕ τελευταία υπάρχει η υπόθεση ότι προσπαθήσατε να σιωπήσετε έναν πρώην υπάλληλό σας για πρακτικές της διοίκησης ε, της τράπεζας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Και για τους δυο σας. Ποια είναι η σχέση της κλασικής τραπεζικής ε, και των επενδυτικών τραπεζών με τους φορολογικούς ε, παραδείσους. Δηλαδή, ποια ε, αξία δημιουργείται εκεί πέρα, πόσους υπαλλήλου ε, έχετε σε φορολογικούς παραδείσους και ποιο είναι το κέρδος εκεί. Ευχαριστώ. Εκτός. Ε, σε παγκόσμιο επίπεδο η UPS έχει πολιτική για την προστασία των ε, καταγγελόντων. Ε, οπότε θα αντέβαινε αυτό σε αυτή την πολιτική. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση τώρα που σχολιάζεται είναι ενεξελίξη η νομική διαφορά οπότε μπορεί αυτό να αποβεί, ό,τι πω εγώ, να αποβεί επιζήμιο για την υπόθεση και άρα δεν μπορώ να το σχολιάσω για το θέμα το, της επενδυτικής και λιανικής ε, τραπεζικής ε, στους φορολογικούς παραδείσους θα σας έλεγα ότι ε, περιοριζόμαστε στην Ελβετία ως προς τη λιανική τραπεζική. Οπότε 0% αυτών των δραστηριοτήτων ελαμβάνουν χώρο σε, φορολογικές, σε φορολογικούς παραδείσους για την επενδυτική τραπεζική. η έδρα είναι στο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό κέντρο του κόσμου, όπου έχουμε με ε, μεγάλες ομάδες ε, ε, πολύ καλά καταρτισμένων ανθρώπων που διευθύνουν αυτές τις επιχειρήσεις. Σε σχέση τώρα με τις, τους φορολογικούς παραδείσους, δεν πρόκειται για προνόμια που προσφέρει ο φορολογικός παράδεισος, αλλά επειδή είτε έχουμε εργαζόμενους εκεί που στο Λουξεμβούργο παραδείγματος χάρη, όπου έχουμε ε, μεσητεία και διαχείριση. 500 υπαλλήλου έχουμε που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και έτσι ε, είναι η αυτή είναι η δομή της αγοράς. Ε, τα νησιά χέιμα χρησιμοποιούνται για hedge funds ή για ε, άλλες υπηρεσίες αντιστάθμισης προς για ε, ε, άλλες υπηρεσίες συγγνώμη, που προσφέρονται στους καταναλωτές, στους πελάτες. Ευελίνα, έχετε άλλες ερωτήσεις? Όχι. Απάντηση Unicredit. Θα είμαι σύντομος. Δεν γνωρίζω ούτε για την Λιαδινική ούτε για την Επενδυτική Πεζική δραστηριότητα σε φορολογικού παραδείσους. Ε, έχουμε μια ε, παρουσία σε αυτούς του επωνομαζόμενου φορολογικούς παραδείσους, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι σε αυτή την ε, Ιταλική εταιρεία holding όλα τα προϊόντα πρέπει να φορολογηθούν στην Ιταλία. Εάν υπήρχε τέτοια χρήση για, τις για τους φορολογικούς παραδείσους, αν υπάρχει, ξαναλέω, Ε, οι φορολόγοι θα ήταν στην Ιταλία. Ε, και όταν χρησιμοποιούμε τέτοια χρηματοπιστωτικά κέντρα σε υπονομαζόμενους φορολογικούς παραδείσους, αυτό γίνεται για καθαρά οικονομικού και επιχειρηματικού λόγου. Σα ευχαριστούμε. Η Σιλβί Γκουλάρ για τους ε, φιλελεύθερου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Σα ευχαριστώ και του δύο που ήρθατε. Δύο ερωτήσει έχω. Η πρώτη ίσω σα ξαφνιάσει. Ε, τι γίνεται στις τράπεζες σας ε, ως προς την ε, έδρα, ως προς την υπηκότητα αν θέλετε. Δηλαδή μας λένε αυτή είναι γαλλική, αυτή είναι ιταλική τράπεζα και τελικά συνειδητοποιούμε ότι είστε διασυνοριακοί. και όταν σας βολεύει πάτε και τοποθετείτε τις δραστηριότητες σας στο σημείο που σας βολεύει περισσότερο. Οπότε... Δεν είναι απαραίτητα εύκολο το ερώτημά μου. Πιστεύετε ότι είστε Ελβετός ή Ιταλός γιατί εκείνη η έδρα ε, της εταιρείας σας ε, ε, ή συνεχίζετε αυτή την διασυνοριακή αλήθεια χωρίς καν να αναρωτιέστε. Και δεύτερον, Α, θα αλλάξει τίποτα με την νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα, θα πάτε τι υπηρεσίε σα στο Λονδίνο, παραδείγματο χάρη, να αλλάξει νομοθεσία ή θα παραμείνετε εσεί στην κυρία Ήπειρο. Η Ιταλία θα απαντήσει ναι, το ίδιο ερώτημα και για τους δύο. Θα μας τα πείτε Ιταλικά. Είμαι περήφανος που είμαι Ιταλός. Μπορείτε να τα πείτε στα Ιταλικά. Η Σιλβί Γκουλάρ μιλάει Ιταλικά. Αισθάνομαι πολύ περήφανος που είμαι Ιταλός. Πιστεύω πως ε, το καθήκον ενός διευθυντικού διευθυντή είναι να εφαρμόσει κατά γράμμα την νομοθεσία εκεί όπου ε, δραστηριοποιείται ο όμιλος και ακριβώς αυτό είναι ο σεβασμός του νόμου και γι' αυτό και θεωρώ πως ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εναρμονισής είναι ο καλύτερος τρόπος για να ε, επιτευχθεί αυτό. Όσον αφορά τα περί Brexit, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος και μπορώ να δώσω μια απάντηση σε σχέση με αυτά που λέμε στην Ιταλία και ως ε, καλός ε, οικογενειάρχης που λέμε στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν αυτό θα οδηγήσει σε μετακινήσεις εταιριών. Εγώ ως Ιταλός και ως Ευρωπαίος θεωρώ πως αυτό θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα και κατά συνέπεια μπορώ να φανταστώ ότι όπως πάντοτε όταν υπάρχουν ε, κρίσεις υπάρχουν και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αλλά αυτό δεν το εύχομαι. Εύχομαι ωστόσο να υπάρχουν σαφείς κανόνες ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να προοδεύσουμε. Ευχαριστώ και εγώ σας σας ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά σε προσωπική μου άποψη μπορώ να σας πω, ε, δεν έχουμε πολιτική ο UBS. Είμαστε Ελβετοί και πολυεθνικοί. Είμαστε Ελβετοί ε, από λόγω κληρονομιάς, γιατί εκεί άρχισε να λειτουργεί ο όμιλος. Ε, για να μπορούμε όμως να εξυπηρετήσουμε αποτελεσματικά τους πελάτες μας πρέπει να είμαστε πολυεθνικοί. Προς το, αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πελατών μας. Στη σήμερα ημέρα ο κόσμος μικραίνει και για να μπορεί μια τράπεζα να εξυπηρετεί ε, καταλήλως την πελατεία της πρέπει να είναι πολυεθνική. Τώρα όσον αφορά το Brexit είναι πολύ περίπλοκη κατάσταση και υπάρχουν πολλοί που ανησυχούν για τις επιπτώσεις του, όχι μόνο για την Ένωση αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Και στο βαθμό που η UBS έχει αντίδραση θα εξαρτηθεί αυτό από τα στοιχεία και τις περιστάσεις συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσο θα υπάρξει Brexit ή όχι. Και όταν αυτά θα αξιολογηθούν τότε θα λάβουμε αποφάσεις. Από την άλλη πλευρά, θα, αν υπάρξει αυτή η καταστροφή, θα προσπαθήσουμε να αντισταθμίσουμε την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου με την είσοδο της Ελβετίας. Χαριτολογεί ο Πρόεδρος και τώρα ο Φάβιο Ντεμάση. Ερώτηση προς την UBS. Επειδή συχνά ταξιδεύω στην Ελβετία, ταξίδευα στην Ελβετία με τη Γερμανίδα γιαγιά μου, θυμάμαι να με ρωτά ένας αυστηρός ε, συνοριοφρουρός να... να μας ρωτά πάντα τι ερχόμαστε να κάνουμε στην Ελβετία και, να δηλω... και αν είχαμε να δηλώσουμε τίποτα. Η γιαγιά μου πάντα, επειδή ήταν πολύ συντηρητική, έλεγε τι... γιατί πηγαίναμε και γιατί όχι. Εσείς τώρα έχετε εξελιχθεί, έχετε δραστηριότητες σε πάνω από 40 χώρες. Και βλέπω την έκθεσή σας για το 2014 και την αναχω... τις αναχώρα εκθέσεις. Οι δημοσιεύσεις σας ε, in scope, όπως ε, δημοσιεύονται και όπως ορίζονται από το CRD4, είναι το μόνο πεδίο εφαρμογής. Ε, αλλά εντός, in, in scope, είναι πραγματικά εφεύρεση αυτή η έννοια. In scope είναι εφεύρεση της ε, UBS. Δεν περιλαμβάνεται πουθενά ε, σύμφωνα με το, και δεν ισχύει σύμφωνα με το 89 της ε, CRD4. Θέλω να γνωρίζω λοιπόν τι ακριβώς σημαίνει. Και έπειτα τα στοιχεία CBC πρέπει να δημοσιεύονται για κάθε κρατοσμένος και για τις τρίτες χώρες όπου έχετε θηγατρικές θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω πόσες θηγατρικές έχετε, ε, Barclays για παράδειγμα, που δεν είναι και αυτή καμιά μικρή εταιρεία, αφού έχει 1329, 1329 παραρτήματα για τα οποία δεν έχουμε καμία απολύτως πληροφορία. Υπάρχουν ένα σωρό είδη καταστημάτων, παραρτημάτων, θηγατρικών που άμεσα ή έμεσα συνδέονται με την μητρική ε, Μια που σε λίγο θα έχουμε αυτές τις νέες διαρροές από τον Παναμά, αναρωτιέμαι αν χρησιμοποιείται trust services εκεί πέρα για άλλου είδους υπηρεσίες για να μπορούν οι ιδιώτες να κρύψουν τον πραγματικό τους πλούτο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά, όσον αφορά την οδηγία CRD4, αυτή αφορά τράπεζες οι οποίες βρίσκονται υπό την αρμοδιότητα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών. Οπότε για τέτοιες ε, τράπεζες πράγματι υποβάλλουμε τις σχετικές εκθέσεις. Επίσης για τις εκθέσεις αναχώρα τις υποβάλλουμε στις ανάλογες ε, φορολογικές αρχές ε, και στην Ελβετία όπως απαιτεί η BEPS και η Ελβετική νομοθεσία. Μπορείτε να μου εξηγήσετε όμως τι είναι το ίνσκο. Και δεν πρέπει να φέρεστε σαν την FIFA γιατί μπορεί αυτό να γυρίσει μπούμεραγκ όπως συνέβη και στην περίπτωση της FIFA. Ναι, δεν ξέρω ποια είναι η ερώτησή σας ακριβώς. Η CRD4 ισχύει για ε, τράπεζες οι οποίες ε, υπόκεινται στον Ευρωπαίο ρυθμιστή. Και άρα δεν ισχύει για την ε, οντότητα που αναφέρατε. Π.χ. έχουμε τράπεζες στις ΗΠΑ, στην Ελβετία, στο Χονγκ Κόνγκ, στη Σιγκαπούρη. Οι τράπεζες αυτές δεν υπόκεινται στις απαιτήσει αυτής της οδηγίας. Ναι, αλλά δεν μας απαιτήσατε. Τι είναι η έννοια scope στις εκθέσεις αναχώρα. Θα έπρεπε νομίζω να απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση. Κοιτάξτε, η έννοια scope για την οδηγία για τις κεφαλαίκες απαιτήσεις, όπως είπα, αφορά μόνο τράπεζες που υπόκεινται στις ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν έχουμε άρα υποβάλει τέτοιες εκθέσεις αναχώρα γιατί δεν απαιτείται. Και για τον Παναμά, δεν γνωρίζω τις δραστηριότητες μας στον Παναμά. Πιθανότατα έχουμε γραφείο εκεί, αλλά δεν το γνωρίζω. Έχετε υπηρεσίες Trust εκεί. Και πάλι σας λέω δεν ξέρω τι υπηρεσίες προσφέρουμε στον Παναμά. Οπότε θα μας στείλετε μια γραπτή απάντηση. Ευχαριστώ. Ε, αν ήμασταν σε δικαστήριο τώρα θα έλεγα ότι δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Euh, λοιπόν, γραπτός θα την πάρουμε την απάντηση. Ο κύριος Φεν Γκίγκολ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα σύντομο ε, ερώτημα προς τη UBS και μετά προς την Unicredit. Πρώτον, UBS. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διάβασα το, την υποβολή στοιχείων για τις εκθέσεις αναχώρα και λέτε εκεί ότι η UBS Limited με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 24 εργαζομένους που έχουν κέρδη 77 εκατομμύρια με φόρο μόνο 3,6%. Πώς τα καταφέρνετε να έχετε τέτοια κερδοφορία ανεργαζόμενο. Και γιατί είναι τόσο χαμηλή η φορολογία. Πώς είναι τόσο ε, ε, ε, αποδοτικοί αυτοί οι άνθρωποι στο Λονδίνο. Γιατί γίνουν credit τώρα. Τα, η υποβολή στοιχείων δείχνει δύο φορολογικούς παραδείσους, Βερμούδες και Κέιμαν. Αν δούμε τον, τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία βλέπουμε και θυγατρικές και στο Χόγκον και στην Τελαουέρ και στο Τζέρζεϊ πέρα από αυτά τα δύο. Μας δίνετε, παρακαλούμε, περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες που έχετε σε αυτές τις δικαιοδοσίες. Και δεύτερον, ξαφνιαστήκαμε όταν ανακαλύψαμε πως τα κέρδη στα, στους, ε, στα είναι διπλάσια από το τζίρο ε, σε σχέση με την, και στην Ιρλανδία τριπλάσια από το τζίρο. Και είναι χαμηλή η φορολογική συντελεστές και στις δύο περιπτώσεις. Είναι Πραγματικά ε, ε, προκαλούν έκπληξη αυτά τα στοιχεία. Μπορείτε να δώσετε κάποιες εξηγήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. UBS πρώτα. Ναι. Η τράπεζα αυτή, η UBS είναι η κύρια επενδυτική μας τράπεζα στον Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει 24 ε, μονίμους υπαλλήλους και άλλους υπαλλήλους από την UBS London το χαμηλός ε, πραγματικός φόρος προκύπτει από το ότι λόγω των αυξημένων προβλέψεων κερδών καταφέραμε να έχουμε κάποιο φορολογικό όφελος ε, το οποίο να αναβάλουμε επίσης την πληρωμή κάποιων φόρων, απλά την αναβάλαμε χρονικά. Ποια είναι η πηγή αυτής της αναβολής. Κοιτάξτε, πρόκειται για ζημίες οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και έχουν μετατοπιστεί χρονικά. Μάλιστα, ε, οι ζημίες από τι προκλήθηκαν ε, δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο, στο υποκατάστημα της UBS AG. Σας ευχαριστώ και διευθυντά της Unicredit. Όπως προσπάθησα να σας εξηγήσω και πριν, η κατάσταση στην Ιταλία είναι κάπως διαφορετική γιατί πρέπει να έχετε κατά νου πως όλα τα κέρδη από τις ε, χώρες που αναφέρατε είναι κέρδη τα οποία είτε φορολογούνται τοπικά στην Ιταλία είτε στο κατάλληλο επίπεδο. Και για να γίνει αυτό πρέπει να κοινοποιήσουμε τις συναλλαγές στις ταλικές φορολογικές αρχές. Οπότε το αποτέλεσμα είναι ότι αν θεωρούν ότι έχει επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο φορολογίας παραμένει η φορολογία σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Ναι, αλλά πρέπει παρόλα αυτά να δηλώνεται αναχώρα. Οπότε, ε, και αν, ακόμα και αν φορολογείτε στην Ιταλία, πρέπει να κάνετε τις δηλώσεις. Ναι, αναφέρεστε σε εκθέσεις αναχώρα σε σχέση με την CRD4. Ενώ από φορολογική σκοπιά, νομίζω πως αυτό θα πρέπει να το δούμε στις εκθέσεις αναχώρα που θα υποβληθούν για την Ιταλία για το 2016 και θα συνταχθεί η εκθέση το 2017. Οπότε έχουμε δύο διαφορετικές εκθέσεις και αυτό δημιουργεί κάποια σύγχυση. Και μπορεί να ρωτήσει κάποιος επενδυτής ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων. Αλλά το δεύτερο σύστημα, το TAX 1, είναι αυτό το οποίο νομίζω απαντά την ερώτησή σας απευθεία. Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου η CRD4 είναι σαφής. Οπότε σας ερωτώ εάν ε, θα διορθώσετε τις εκθέσεις σας και θα μας δώσετε τις ε, πληροφορίες ε, που απαιτεί το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Με συγχωρείτε, δεν είμαι ειδικό στη CRD4, εγώ είμαι ειδικό στα φορολογικά και όπως επεσήμανα, ίσως να μην ήμουν σαφής, τα δεδομένα στα οποία αναφέρεστε δεν είναι φορολογικά δεδομένα είναι ε, δεδομένα που δίδονται για τις ρυθμιστικές αρχές. Οπότε, αν δείτε την φορολογική μας θέση συνολικά, τα κέρδη μας εκεί φορολογούνται πλήρως σύμφωνα με πολύ αυστηρή νομοθεσία, την Ιταλική. Η δεύτερη ερώτηση για τα Cayman και τα κέρδη εκεί και στην Ιρλανδία και αλλού. Κύριε Πρόεδρε, η απάντηση είναι η ίδια. Είμαστε παρόντες εκεί ε, καθαρά για επιχειρηματικούς σκοπούς. Αν έχουμε κέρδη εκεί και σε κάποιες περιπτώσεις ε, δεν έχουμε κέρδη, γιατί είμαστε εκεί παρόντες για επιχειρηματικούς σκοπούς, τότε φορολογείται αυτό το κέρδος σύμφωνα με τους κανόνες που μόλις ανέφερα. Εγώ ρώτησα για την πηγή αυτού του εισοδήματος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο τζίρο. Και μια που έχει τελειώσει ο χρόνος, μπορείτε να μας απαντήσετε γραπτός για να έχουμε μια κανονική απάντηση. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Χίλια ευχαριστώ. Αχα, θα στείλετε γραπτό την απάντηση. Ο Μάρκο Τσάνι για το ευθύτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση προς την οποία αφορά την πρόσφατη καταδίκη των Βρετανικών αρχών για ορισμένα σχέδια που χρησιμοποιούσε η UBS και άλλες τράπεζες για να αποφύγουν τις φόρους επί των μπόνους, επί των πριμ των διευθυντών τους, των μάνατζερ τους. Αυτό γινόταν μέσω της απόδοσης μετοχών εταιριών που είχαν δημιουργηθεί ακριβώς για να αποφευθεί η φορολογία επί αυτών των μπόνους ο δικαστής που εξέδωσε την απόφαση ε, ανέφερε και παραθέτω. Είναι τα πιο σύνθετα σχέδια που έχουν ποτέ φτιαχτεί για να αποφευχθούν οι φόροι. Υπάρχει μεγάλη δαπάνη πνευματικής ε, ενέργειας για να που αφιερώνεται στην αποφυγή της φορολογίας. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν ποια είναι η αξιοπιστία των τραπεζών που όπως εσείς ε, σήμερα έρχεστε εδώ και δικαιολογείτε αυτές τις περίπλοκες οργανωτικές δομές ε, και που χρησιμοποιούν τη φορολογική παράδειση αποκλειστικά έτσι ώστε να παρακάμψουν ρυθμίσεις και να αποφύγουν την καταβολή φόρων. Και η ερώτησή μου για τον εκπρόσωπο της Unicredit είναι η υπόθεση της επιχείρησης Brontos. Πρόκειτο σύντομα για μια περίπλοκη χρηματοπιστωτική δομή ανάμεσα στην Ιταλία και το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο που με ένα παιχνίδι εικονικών μεταεμβασμάτων σε τουρκικές λίρες μάλιστα γινόταν διάφορες συναλλαγές για να ε, αποφευθούν ε, οι φόροι. Πρόκειται για αποφυγή 264 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά προχώρησε η διοικητική διαδικασία και υπήρξε μία λύση. Θα ήθελα ένα σχόλιο λοιπόν για αυτές τις συμφωνίες από πλευρά σας. Ε, εσείς δεν πιστεύετε πως αυτά αντιστοιχούν σε ένα είδος... Ε, φοροδιαφυγής και δεν αποθαρρύνατε αυτές τις διαδικασίες ε, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι χαμηλότερο το τελικό αποτέλεσμα ε, από ό,τι θα καταβαλόταν αρχικά. Τέτοιου είδους δηλαδή φοροδιαφυγές αποφεύγονται με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ κύριο Σπίνιο, χωρίς μικρόφωνο. Μιλάμε για, εδώ για ερμηνεία ένα πολύ τεχνική φύση ε, σημείο. Πρόκειται για ένα σχέδιο κεφαλοποίηση από το 2003. Εμεί ε, έχουμε απογοητευθεί με, από το αποτέλεσμα, αλλά καλωσορίζουμε την προσοχή που έδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πολιτιστικέ ε, προδιαγραφέ ανάλογα με την φορολογία διαφέρουν. Πριν από 20 χρόνια όλοι κάπνιζαν στα εστιατόρια και στα μπάρα. και η φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο καθοδηγείται αποκλειστικά από συγκεκριμένο τύπο. Από τη στιγμή που κανείς τύπη συνεντάξει μπορεί να ρυθμίσει όπως θέλει τα πράγματα με στόχο να μειώσει την φορολογία. Όπως και το κάπνισμα στα μπαρ πλέον αυτό δεν είναι αποδεκτό και η UBS έχει προσαρμόσει τις πρακτικές της αντιστοίχως. Μια τυχές που μια υπόθεση που χρονολογείται πριν από 14 χρόνια αποφασίστηκε φέτος, αλλά έτσι λειτουργεί η νομοθεσία σε πολλές δικαιοδοσίες. Άρα λοιπόν αυτές οι πρακτικές ε, δεν ισχύουν πλέον εδώ και 14 χρόνια, λέει ο Πρόεδρος. Από την άποψη της UBS, ναι, μία φορά το κάναμε το 2013 λέει ο μιλητής και δεν το έχουμε επαναλάβει, μάλλον το 2003. Μάλιστα, ευχαριστώ Credit για λόγους ευγένειας ε, σε... απέναντι στον συμπατριώτη μου Ιταλό θα μιλήσω στα Ιταλικά. Θα ήθελα καταρχάς να αποσαφηνίσω ένα σημείο. Η υποτιθέμενη συναλλαγή Μπρόντος είναι μια πολύ περίπλοκη συναλλαγή που ήταν όμω κοινή ως, τύπος, τυπολογία σε μια περίοδο της ιστορίας μας και όσον αφορά την προστασία των θεσμών, των χρηματοπιστωτικών θεσμών. Αυτή η επιχείρηση έγινε σε μια φάση ερμηνείας που δόθηκε από πρωταρχικές μελέτες σε, πολλές, σε πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το σημαντικό στοιχείο πέρα από το γεγονός ότι η Ιταλική Φορολογική Αρχή δεν το χαρακτήρισε ήταν ότι το γεγονός ότι η Unicredit τότε έκανε αυτή την επιχείρηση με καλή πίστη και με πλήρη διαφάνεια, υποδεικνύοντας μάλιστα ρητά σε όλα τα τεκμήρια, σε όλα τα έγγραφα και μάλιστα τη στιγμή που η αρμόδια δημοσιονομική αρχή εξέφρασε αμφιβολίες ενημερώσαμε την λόγω αρχή γιατί μας ζήτησε μια εξήγηση αλλά έδωσε μια ε, ερμηνεία διαφορετική σε σχέση με τα στοιχεία της Unicredit. Όλα αυτά που σωστά υπογραμμίσατε αποδείχθηκαν κιόλας από την τελική απόφαση του ανώτατου Ιταλικού εφετείου που αναγνώρισε ότι δεν υπήρχε καμία ε, ένοχη ή ε, ε, ζημιογόνα δράση από πλευρά τη Γενική. Κατά συνέπεια, δέχομαι το γεγονό ότι μπορεί να δοθούν διάφορε ερμηνείε, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση, το γεγονος οτι μπορει να δοθουν διαφορες ερμηνειες αλλα αυτή του αποχαρακτηρισμού μιας πολύ περίπλοκης διαδικασίας ε, είναι ένα είδος έγκρισης ή συγκατάθεσης. Πρόκειται για μια διαδικασία ανάμεσα σε μια διοίκηση και έναν φορολογούμενο που ασκεί πολύ περίπλοκες διαδικασίες. Το να σκεφτεί κανείς διαφορετικά θα σήμερα ότι εμφισβητεί το γεγονός ότι η Ιταλική εφορία ε, φάρμοσε σωστά τους νόμους, πράγμα το οποίο οφείλει να κάνει. Ε, ναι, Μπερνάρ Μονό από την ΕΝΕΦ. Ευχαριστώ. Εγώ απευθύνομαι στην ΕΜΠΕΣ. Ευχαριστώ τον κύριο Πίνο που είναι παρόν. Αν χρειαζόταν να κάνουμε ένα παλμαρέ των όσων δείχνουν περισσότερο κινησμό, ε, θα ανέφερα τέσσερι τράπεζε παγκόσμιε. Ε, ο JP Morgan, ο βασικό ένοχο ε, τη κρίση στο subprime το 2007, Goldman Sachs για το 2001, η Και τέλος ε, η τελευταία είναι η UPS για το ρόλο της ε, στην, στην φοροδιαφυγή των ε, ιδιωτών. Το 2013 ήσασταν πρώτοι στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Για να το κάνετε αυτό έχετε φτιάξει ένα επιθετικό σύστημα για τους πλούσιους πελάτες σα, ώστε να τους κάνετε να ανοίξουν έναν μη δηλωμένο λογαριασμό κυρίω στην Ελβετία. Στη Γαλλία έχετε διωχθεί δικαστικά για φοροδιαφυγή. Το 2008 υπήρχαν 38.000 ε, λογαριασμοί για ένα ποσό των 4 δις ε, ενεργητικού. Έχετε πάψει αυτές τις αθέμητες πρακτικές ε, για να αναγκάσετε τους πελάτες σας να ανοίγουν λογαριασμούς και offshore. Ποιες είναι οι ποινικέ και διοικητικές διαδικασίες εναντίον σας αυτή τη στιγμή στον κόσμο και έπειτα τι ακριβώς συμβαίνει όσον αφορά τις φορολογικές καταδίκες στην Γαλλία. Ναι, εδώ μιλάμε για την φορολόγηση των πολυεθνικών εταιριών. Αυτό είναι η ακρόασή μας. Παρακαλώ, κύριε Πίνιο. Σχετίζονται όλα αυτά με την ιδιωτική τραπεζική ε, και τα θέματα της ε, μεταφοράς ε, στοιχείων ενεργητικού και δεν υπάρξαν τέτοιες αθέμητες πρακτικές για να χρησιμοποιήσουμε την Ελβετία ως μηχανισμό για να συμβάλλουμε στη φοροδιαφύγη και φοροαποφυγή. Έχουμε διάφορες συμφωνίες με δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο που ενισχύουν τη διαφάνεια υπέρ αυτού, ε, αυτών των οργάνων που ισχύουν για τις υπόλοιπες ε, ε, τράπεζες. Η ΦΑΤΚΟ παραδείγματος χάρη για τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων, τον είπαμε. Χρειάζομαστε θετική δήλωση για τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, ε, είτε μιλάμε για τα, ε, τις οντότητες είτε για τους πελάτες. Ε, και πάντα ενθαρρύνουμε τους πελάτες ενθελουσίως να δίνουν πληροφορίες σε σχέση με την φορολόγηση των καταθέσεων. Τούτου λεχθέντος έχουμε μάθει πάρα πολλά επώδυνα και όλες από αυτό τον κώδικα διοντολογίας. Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση από φορολογικής πλευράς να κάνουμε το σωστό. Και μας βοηθούν οι κανόνες που έχουμε, δεν θα ε, συμβάλλουμε σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, ούτε και θα βοηθήσουμε τους πελάτες μας να το κάνουν. Και σε σχέση με τις άλλες δύο ερωτήσεις για τη Γαλλία, ε, ε, είναι προϊούσα διαδικασία και δεν ε, είμαι εξουσιοδοτημένος να το σχολιάσω γιατί ενδεχομένως οι δηλώσει μου να αποβούν επιζήμιες ε, στα πλαίσια αυτής της ε, νομικής διαδικασίας. Ο κύριος Μονό. Ναι, κύριε Πινό, όμω δεν απαντήσατε για τι ποινικέ και διοικητικέ διαδικασίε ανά τον κόσμο. Πέραν της Γαλλία, υπάρχουν και αλλού. Είπα, δεν μπορώ να σχολιάσω όταν είναι μια υπόθεση ποινική ή άλλη εν εξελίξη. Ζητώ συγγνώμη, δεν είμαι εξουσιοδοτημένος να απαντήσω. Πρόεδρος, διαχωρισμός νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας. Ε, ε, ο κύριος Μπάλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, όπως ήδη είπαμε θα ήθελα να απευθυνθώ στον εκπρόσωπο της ε, Unicredit και να θέσω ένα ερώτημα που είναι και κάπως γενικότερο. Πρώτα απ' όλα, διάβασα και είχα ακούσει και στο παρελθόν πως ε, πριν από λίγους μήνες σε μια δίκη στη Γερμανία στην, ε, σε, σε περιπτώσεις COMEX καταδικαστήκατε σε ένα πρόστιμο 30 εκατομμυρίων ευρώ. Να δεχτούμε μια τέτοια σύγκριση υπάρχει νομίζω μια υποψία ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία τρέχουν εδώ, τα οποία δεν θα θέλατε ε, να βγουν δημοσίως. Το ερώτημά μου λοιπόν, ε, όλα αυτά γύρω από την περίπτωση COMEX, ε, πώς αφορούν την Hippo Bank, την γερμανική θηγατρική σας και αν έχουν τελειώσει αυτές οι περιπτώσεις. Και κάτι άλλο το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, ποιο ρόλο συνολικά παίζουν τα φορολογικά μοντέλα για να προσελκύσετε μεγάλους πελάτες. Ιδιαίτερα πελάτες ιδιαίτερης οικονομικής επιφάνειας. Κάποιοι εύποροι πελάτες θα μπορούσαν, υποφελούνται από τέτοια φορολογικά μοντέλα ή όχι. Merci, Monsieur le Thank... Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις που εκκρεμούν ακόμα στα δικαστήρια, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω. Θα προσπαθήσω να απαντήσω χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες που δεν πρέπει. Πόσο κατάλαβα να φέρεστε σε συναλλαγές που έγιναν από το 2005 μέχρι το 2008. Οπότε μιλάμε για το παρελθόν. Θα ήθελα να απαντήσω λοιπόν στην δεύτερη ερώτηση. Έχουμε και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ε, ένα πολύ στιβαρό πλαίσιο φορολογικής συμμόρφωσης και τοπικά και στη Γερμανία και παγκοσμίω. Τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση την οποία δεν μου επιτρέπεται να σχολιάσω θα ήθελα να επισημάνω ότι ε, στη Γερμανία και οπουδήποτε αλλού γνωρίζω σε θελοντική βάση παρουσιάζουμε τα όσα ξέρουμε στις φορολογικές αρχές και ζητάμε την καθοδήγησή τους γιατί σκοπεύουμε να είμαστε όσο να τον πιο διάφανοι. Οπότε στις περιπτώσεις αυτές, από όσο γνωρίζω, υπήρχε ένα αίτημα πλήρους διαφανής από τη δικιά μας την πλευρά πριν ε, απευθυνθούν σε εμάς οι αρχές. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Μπορκχαρτ. Εν μέρη ρώτησα μετά μια που είμαστε τόσο μια που είστε τόσο ανοιχτοί και συνεργάσιμοι με τις αρχές έχετε αυτό το πρόστιμο των 30 εκατομμυρίων ευρώ και ακόμα δεν έχουν κλείσει όλες οι περιπτώσεις αυτό σημαίνει πως μάλλον δεν θέλετε περισσότερη δημοσιότητα για αυτές τις ε, περιπτώσεις. Ε, δεν ξέρω, μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό. Δεν γνωρίζω κάποια συγκεκριμένη πληρωμή 30 εκατομμυρίων. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι όταν καταλήγουμε σε ένα συμβιβασμό με τις ε, φορολογικές αρχές θα το κάνουμε για να συμμορφωθούμε. Όχι για λόγους δημοσιότητας ή μη δημοσιότητας. Ναι, μια που κάποιο σας ενημέρωσε ή η εφημερίδες ή δεν ξέρω πω. Ε, προφανώς υπάρχει δημοσιότητα. Οπότε το θέμα δεν είναι ότι θέλουμε να αποφύγουμε τη δημοσιότητα, θέλουμε να συμβαστούμε και να διορθώσουμε ένα λάθος. Δεν ήταν οι φορολογικές αρχές, ήταν το δικαστήριο αυτό το οποίο σας επέβαλε το πρόστιμο στην κολονία γνωρίζετε πως υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες σε διαφορετικές χώρες. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν ε, ποινές από τις φορολογικές αρχές, σε άλλες χώρες υπάρχει λεγόμενη αποζημίωση για να ανακτηθούν τα κέρδη. Αυτό είναι ένας κανόνας που υπάρχει στη Γερμανία. Οπότε, όπως σας είπα, δεν μπορώ να συζητήσω αυτή την υπόθεση, αλλά αν μιλάτε για τέτοια ε, περίπτωση είναι κάτι το φυσιολογικό. Υπάρχουν ε, και πολύ χαμηλά πρόστιμα και πιθανή ανάκτηση των κερδών. Είναι ένας γερμανικός κανόνος. Ε, δεν είμαι ειδικό στο γερμανικό φρολικό δίκαιο, πιθανώς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Σας ευχαριστώ. Sí, yo quería hacer dos preguntas. Θέλω να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις προ την ε, τράπεζα UBS, ε, τον κύριο Πινιό. Η πρώτη είναι, μήπως μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε ότι ως συνέπεια μιας ε, έρευνας που έκαναν η ΕΠΑ για τη δική σας τράπεζα το 2008, χρειάστηκε να καταβάλλεται ένα πρόσημα 730 εκατομμυρίων δολαρίων σε μεγάλο μέρος ως ερευνά που προέκυψε για να βοηθηθούν ε, κάποιοι πολίτες να αποφύγουν τη φορολογία. Άκουσα την προηγούμενη σας απάντηση κύριε Πινιό ότι η UBS σταμάτησε το κάπνισμα για να συνεννοιόμαστε. Δηλαδή έμαθε πολύ καλά τα μαθήματα, τα διδάγματα και σας πιστεύω. Όμως τότε διερωτώ με και ακριβώς σας ρωτώ και εσάς γιατί για το ίδιο πράγμα, το ίδιο, την ίδια κατηγορία, δηλαδή τη δυνατότητα να οι, μεγάλοι πελάτες με μεγάλες περιουσίες να αποφευγούν την φορολογία. Γιατί λοιπόν σας, έχουν, σας διώκουν ποινικά η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο το 2012 με 2014. Μπορείτε να μου επιβεβαιώσετε αν ισχύει αυτό ή όχι. Και κατά δεύτερο λόγο, οι ΕΠΑ ξεκίνησαν για την UBS ε, μια δικαστική έρευνα μόλις το Φεβρουάριο του 2015, πριν ένα χρόνο δηλαδή, ε, και αναφέρονται στα bearer bonds για το το, τα ομόλογα του στον κομιστή είναι μια πρακτική, ένα προϊόν ε, ε, οικονομικό συμβατό με αυτά που είπατε και εγώ συμμερίζομαι, βέβαια συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να είναι αυτός ο στόχος, ότι δηλαδή η τράπεζα να έχει μια βιώσιμη αξία μακροπρόθεσμα, δηλαδή ε, μπορεί η έρευνα αυτή για τα ομόλογα του κομιστή να μπορεί αυτή να οδηγήσει σε νέα κύρωση ποινή για την τράπεζά σας και εάν υπάρχει κάποιο είδος μια υπηρεσία εσωτερικής ε, αστυνομίας, εποπτείας, ελέγχου μέσα στην τράπεζα, ώστε οι δραστηριότητε των πελατών της τράπεζάς σας ε, να μην καταλήγουν ε, στο να σχετίζονται με την φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή. Υπάρχει κάποιο σύστημα εσωτερικό για την εποπτεία. Ευχαριστώ. Yes, I can confirm as is part of the public record that in ε, Θέλω να σας πω ότι για το 2008-2009 για τα πρακτικά έκανε μια συμφωνία με την εισαγγελία των ΗΠΑ σε σχέση με την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών από την Ελβετία προς τις ΗΠΑ για την ε, πώληση χρεογράφων και την ε, παροχή ε, συμβουλών για φοροαποφυγή, διότι είναι θέμα ποινικού και όχι αστικού δικαίου για τους πελάτες στη ΣΥΠΑ. Πέραν αυτού δεν υπέβαλαν ε, τις ε, σχετικές ε, δηλώσεις ως προς αλλοδαπούς λογαριασμούς. Για τις υπόλοιπες χώρες δεν ξέρω να υπάρχουν άλλες ε, διαδικασίες εν εξελίξη για τη Γερμανία. Ολοκληρώθηκε το 2014 μια διαδικασία. Πληρώσαμε 300 δίσε σε πρόστιμα και ανάκτηση ποσών ε, στη γερμανική κυβέρνηση για αντίστοιχες ε, διασυνοριακές καταστάσεις ανάμεσα στην Ελβετία και τη Γερμανία. Για τη Γαλλία και το Βέλγιο, ξαναλέω, είναι προϊούσες οι διαδικασίες, δεν εξουσιοδοτούμε να τα σχολιάσω. Για το δεύτερο ερώτημα για τα ομόλογα στον κομιστή. Δεν ε, μπορώ και πάλι να σχολιάσω διαδικασίες εν εξελίξη. Θα έλεγα όμως ότι αυτά τα ομόλογα είναι επικίνδυνα διότι είναι ομόλογα στον πραγματικό κομιστή που είναι εξαιρετικά σπάνια βάση του τωρινού χρηματοπιστωτικού συστήματος οπότε κάποιος ε, φορολογούμενος αμιλητός ε, μπορεί να ε, αποκομίσει ένα κέρδος που πολύ δύσκολα μπορεί να εντοπίσει μια φορολογική αρχή. Εμείς συμφωνόμαστε με ε, την κείμενη νομοθεσία για, τις, ε, για τα ομόλογα στον κομιστή. Αλλά το θέμα είναι ότι στην ουσία παγκοσμίω ε, δεν υπάρχουν πλέον ουσιαστικά ομόλογα στον κομιστή. Πρόκειται για καταχωρισμένα χρεόγραφα στην ουσία. Ευχαριστούμε. Ο Διευθυντής της Unicredit. όχι και πάλι όχι. Το αντίθετο. Ε, ε, στη συμμόρφωση ε, έχουμε πολύ καλές επιδόσεις. Η σχετική υπηρεσία εντοπίζει τα λάθη και ό,τι εντοπίζει αυτά που δεν είναι αποδεκτά βάσει του κώδικα δεοντολογίας. Και γιατί κάνουμε τη διερεύνηση, διότι θέλουμε να επιτύχουμε την συμμόρφωση ε, ανάλογα με τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχουμε. Ευχαριστούμε. Κλείσαμε το τρίτο πάνελ. Θα ήθελα να αντλήσουν τα συμπεράσματα ε, οι δύο συνεισηγητές μας από τις τρεις ε, ακροάσεις αυτού του απογεύματος, Κόφωτ και το Έρερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους εκπροσώπους των τραπεζών για την παρουσία τους. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση μας σήμερα δείχνει ότι οι εκθέσεις ε, αναχώρα που είναι πια υποχρέωση για τις τράπεζες είναι πάρα πολύ χρήσιμες γιατί αποκαλύπτουν κάποια από τα προβλήματα του παρελθόντος που υπάρχουν ακόμα και βεβαίω η ανταλλαγή των πληροφοριών που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά δεύτερον, ο ρόλος μας ως Επιτροπή είναι να εστιάσουμε στο πώς ο χρηματοπιστωτικός τομέας και οι τράπεζες διευκολύνουν την φοροαποφυγή των επιχειρήσεων και εκεί πέρα νομίζω πως έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε Λάμαντα, υπόψη πως ε, σήμερα πλούτος που βρίσκεται στο offshore είναι στα 13 εκατομμύρια δολάρια είπα και το 1 τρίτο των ε, εταιρικών επενδύσεων περνάνε μέσα από υπεράκτιες ε, επικράτειες και γνωρίζουμε πως 72% της μεταφοράς κερδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μέσω transfer pricing σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οπότε τα νούμερα μας δείχνουν πως υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα εδώ πέρα. Οπότε θα ήθελα να πω πως ε, απαιτείται περισσότερη διαφάνεια και απλούστευση. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεύτερον, θα ήθελα επίσης να πω πως σημαντικός είναι και ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ όλων των ε, εν λόγω δικαιοδοσιών ε, και των δικαιοδοσιών όπου δραστηριοποιείται μια τράπεζα και στους G20 και στον ΩΣΑ αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε λοιπόν σήμερα πως οι τράπεζες ε, αντιμετωπίζουν περισσότερους ελέγχους και έχουν βοηθήσει εδώ πέρα οι εκθέσεις αναχώρα αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και εγώ αναμένω περαιτέρω δουλειά επί των συστάσεων αυτών και τέλος να πω πως ήταν χρήσιμο για μένα το ότι ακούσαμε το ότι οι τράπεζες ε, σε γενικές γραμμές ε, στηρίζουν τις δημόσιες εκθέσεις αναχώρα για τον κλάδο τους και ελπίζω να ισχύσει αυτό για όλους τους ε, κλάδους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Μιχαήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των τραπεζών που ήταν εδώ πέρα και μας απάντησαν, εξαρτήτως του πώς αξιολογεί κανείς τις ε, απαντήσεις. Οπωσδήποτε σε κάποια απάντηση θα θέλαμε μια... σε, κάποια... σε κάποιες ερωτήσεις θα θέλαμε διαφορετικές απαντήσεις ή πιο λεπτομερείς. ή ναι, θα θέλαμε να λάβουμε πληροφορίες ε, για αυτά τα οποία αρνήθηκαν ε, να απαντήσουν οι πρόσωποι λέγοντας πως εκκρεμούν ε, διαδικασίες, αλλά προφανώς πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθούν κάποιες ερευνητικές διαδικασίες για εμάς. Επίσης είναι ενδιαφέρουσες ε, οι ερωτήσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν στην δουλειά της Επιτροπής μας. Σημείωσα πως κάποιοι πρόσωποι είπαν πως ε, η φορολογική γίνεται εκεί όπου δημιουργείται η αξία. Εδώ πέρα λοιπόν τίθεται το ερώτημα του εάν ε, υπάρχουν κάποιες γενικά, γενικά επαρκώς αναγνωρισμένοι ορισμοί για την δημιουργία αυτής της αξίας. Και βεβαίως δεν απαντήθηκε το θέμα της ε, τόσο διαφορετικής παραγωγικότητας στην Ιρλανδία, παραδείγματο χάρη και διαφόρων άλλων τοποθεσιών ε, υπεράκτιων. Και θα πρέπει εδώ να δούμε γιατί σε κάποιους φορολογικούς παραδείσους ε, δημιουργείται τόσο περισσότερη αξία και αν αυτό είναι τελείως ανεξάρτητο από τη φορολογική νομοθεσία. Νομίζω πως θα πρέπει να θεμελιωθεί περισσότερο αυτό το θέμα. Επίσης, Νομίζω ήταν λογικό το ότι ήρθαν εδώ εκπρόσωποι των τραπεζών και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρωτού αντλήσω και εγώ κάποια συμπεράσματα, να υπενθυμίσω πως ε, πριν από το τρίτο πάνελ, ο κύριος Τσεκάτσι θα πρέπει να μας ε, στείλει μια γραπτή απάντηση για το ερώτημα του κύριου Γκίγκολ σε σχέση με ε, το κέρδος ε, και τζίρο και την αναλογία προς τους φόρους για κάποιες οντότητες μη συνεργατικές. Βερμούδες, Κάιμαν και τέτοια. Ιρλανδία. Θα τη θυμάστε την ερώτηση σίγουρα. Και δεσμευτήκατε να μας στείλετε γραπτό στην απάντηση. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τους προσκεκλημένους. Ξέρουμε ότι κλειδονίστηκε και το ε, τραπεζικό περιβάλλον μετά τους Lehman Brothers ε, και εμπλουτίστηκε η νομοθεσία ήταν μεγάλη εξάλλου και συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, προληπτική εποπτεία, παραδείγματο χάρη για την, ε, τον ε, ενιαίο μηχανισμό εποπτείας, σε τα τεστ κοπόσεως που υφίστανται τακτικά οι οντότητες των ομίλων σας οι εξοεδαφικές ε, νομοθεσίες ε, τον ΗΠΑ ε, επίσης μετεξελίχθηκαν. Η ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων ε, που με ιδιαίτερα θεαματικό τρόπο ε, επηρεάζει τις δραστηριότητές σας και κατόπιν πρόοδος ως προς τη διαφάνεια του ίσους όρους ανταγωνισμού, κατάργηση του τραπεζικού απορρίτου. Η UBS έκανε αυτή την παρομοίωση προηγουμένως με την απαγόρευση καπνίσματος σε δημοσίους χώρους. Λοιπόν, εξέλιψε το τραπεζικό απόρριτο με εξίσου ε, απρόσμενο τρόπο όπως και η δυνατότητα καπνίσματος σε δημόσιο χώρο. Ε, στη συνέχεια ένα άλλο στοιχείο του νέου περιβάλλοντος είναι οι εκθέσεις αναχώρα και σήμερα διαπιστώσαμε αφενός ε, το ε, όφελο στις πληροφορίες που αποκτούμε χάρη σε αυτές τις εκθέσεις αναχώρα, ταυτόχρονα όμως το πόσο σημαντικό είναι για μας να ξέρουμε ότι μετά από δύο-τρία χρόνια τελικά μια χαρά ε, προσαρμόστηκαν οι τράπεζες. Αυτή είναι ισχυρότατη επιχειρηματολογία για να αιτιολογήσουμε εφαρμογή του ίδιου συστήματος για όλες τις υπόλοιπες πολυεθνικές. Αυτή τη στιγμή. Ο τόσο ευαίσθητος τομέας τραπεζικής προσαρμόστηκε μια χαρά. Για τις τράπεζες αυτό που καταλαβαίνουμε και για τις δραστηριότητες των πολυεθνικών ε, για, υπήρξε το πριν και μετά τους Lehman Brothers ε, για τις τράπεζες και για τα φορολογικά ζητήματα το ίδιο θα ισχύει με τα Lex Leaks πριν και μετά. Για μας τους νομοθέτες θα πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα από αυτό το σκάνδαλο και οι φορείς ε, της αγοράς πρέπει να λάβουν υπόψη το ότι πλέον Δεν πρόκειται πλέον για φορολογικά τρίκ και τεχνικές. Δεν μπορεί να προσμένουν να, να ε, ε, ελπίζουν σε αυτό το σκληρότατο ανταγωνισμό να επικρατήσουν σε σχέση με ανταγωνιστές και άλλα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με αυτά, με αυτά τα φορολογικά κόλπα. Λοιπόν, ε, έχουμε προβλέψει και άλλες ακροάσεις με άλλες τράπεζες και θα ήθελα ε, να μας στείλετε γραπτός απάντηση. Δεν έχω τίποτα άλλο στην ημερήσια διάταξη, οπότε κυρίζω τη λήξη της συνεδρίασης και τα ξαναλέμε 4 Απριλίου από τις 3 και μετά στις Βρυξέλλες. Ε, θα έχουμε την Επίτροπο Φεστάγκερ για τις νέες πρωτοβουλίες που ανέλαβε ως προς τις χωρικές οι ε, κρατικές συγγνώμη, επιδοτήσεις ε, που θεωρούνται ως ασύμβατες με τη φορολογική νομοθεσία και θα ολοκληρώσουμε και τις ακροάσεις με τους εκπροσώπους της Deutsche Bank και της Royal Bank of Scotland. Σας ευχαριστώ. Λίγη συνεδρίαση.